Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Dear Speaker of the House of Representatives of the Netherlands. Αγαπητέ Πρόεδρε, ΑΡΙΠ της Βουλής των Κοινοτήτων της Ολλανδίας, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Γερουσίας ε, της Ολλανδίας, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή ε, που καλωσορίζω για τη δεύτερη μέρα της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Ομάδας συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια των Κρατών Μελών. Είχαμε χθε τη διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σήμερα έχουμε την διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη ε, για τη σταθερότητα, των οικονομικών συντονισμών και τη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λεγόμενη διάσκεψη του άρθρου 13. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο της ε, Ολλανδίας που συνδιοργανώνει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την εκδήλωση και πρέπει να τονίσω ότι είχαμε συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, το πολιτικό και το διοικητικό, άριστη μάλιστα συνεργασία. Σας ευχαριστώ όπως πάντα με πολύ αποτελεσματικό ολλανδικό τρόπο οργανώσατε αυτή την εκδήλωση. Bedankt für die Generalstaaten. Κυρίες και κύριοι, η οικονομική ανάκαμψη έχει επανέλθει αλλά πολλές προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε το 2016. Η επιβράδυνση της ε, κινέζικης οικονομίας και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες επανεξορρόπησης ε, που περιμένουμε να υπάρξουν με την τιμή του πετρελαίου που εξακολουθεί να είναι χαμηλή και γενικά υπάρχει δραματική κατάρρευση των εισαγωγών από κάποιες αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν επίσης προβλήματα και δεν ανέφερα καν τις γεωπολιτικές προκλήσεις που σίγουρα θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την επικείμενη σε αυτή τη βδομάδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η περίοδος που, είμαι, που, η περίοδος στην οποία ζούμε είναι περίοδος ισχυρών αναταράξεων και όσα γίνονται παγκοσμίω έχουν επιπτώσεις και στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, η κρίση του προσφυγικού, η καταπολέμηση φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η τρομοκρατία κατάσταση με την Ρωσία, την Ουκρανία, η Συρία, η Λιβύη, η κλιματική αλλαγή. Επίσης, το θέμα του υποψηφίσματος παραμονής ή όχι στην Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά δεν είναι θέματα που περάζουν ένα μόνο κράτος μέλος για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ε, προκλήσεις, τις πολυκρίσεις που αντιμετωπίζουμε Πρέπει να επιδείξουμε περισσότερη αλληλεγγύη παρά, ποτέ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεργασία σε επίπεδο ένωσης. Να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα των 530 ε, εκατομμυρίων κατοίκων που έχουμε για να παίξουμε το ρόλο μας στην παγκόσμια σκηνή είναι ο καλύτερος τρόπος για να δράσουμε αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση με βάση τα συμφέροντά μας. Και αν θέλουμε συνεργασία σε ενωσιακό επίπεδο Πρέπει να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού επίπεδου. Η διακοινοβουλευτική συνεργασία παίζει ουσιώδη ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για αυτή τη δυνατότητα να συζητήσουμε με εθνικού βουλευτέ τον οικονομικό συντονισμό και την διακυβέρνηση. Η κρίση τη Ευρωζώνη κατέδειξε τον υψηλό βαθμό αλληλεξάρτηση μεταξύ κρατών που αποφάσισαν ε, να έχουν το ίδιο νόμισμα. Ορισμένα από αυτά χρειάστηκε να διασώσουν άλλα που αντιμετώπισαν υπερβολικό δημόσιο ή ιδιωτικό χρέος και ενισχύθηκε η ενωσιακή συμβολή στις εθνικές οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά τα αλλεπάλληλα μνημόνια και τα σύμφωνα μοιάζει να δημιούργησαν ένα πολιτικό σύστημα ε, που βασίζεται σε ασαφή κατανομή αρμοδιοτήτων. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η αξιόπιστη δέσμευση και η σωστή λογοδοσία σε εθνικό αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξει νομιμοποίηση, το οποίο σημαίνει και δημοκρατική λογοδοσία. Είναι ουσιώδη όλα αυτά για την επιτυχή εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και για αποτελεσματική διακυβέρνηση γενικότερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χθε είχα τη δυνατότητα να μιλήσετε για ένα νέο είδος, είδους ευρωπαϊκό εξάμεινο στο οποίο συμμετέχουν και τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον καθορισμό του κύκλου 2016 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από διάφορες οπτικές γωνίες. Συζητήσατε και τη συνέχεια θα δοθεί ε, στα θέματα τα φορολογικά, στην διάβρωση της φορολογικής βάσης και την προσπάθεια φοροαποφύγης. Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για την δημοσιονομική προσπάθειες συντονισμού για να δούμε πώς το σύμφωνο για τα δημοσιονομικά θα εφαρμοστεί. Χαιρετίζω το γεγονός ότι σήμερα έχουμε την πρώτη διάσκεψη, άρθρο 13, από την έκρηση των ε, διαδικαστικών κανόνων τον ε, παρελθόντα Νοέμβριο. Μετά από πολλά χρόνια. Ε, δυσχερών συζητήσεων. Επιτέλους συζητήσαμε επί μεθόδων εργασίας που θα μας επιτρέψουν να εστιάσουμε πλήρως, όχι πλέον στους κανόνες λειτουργίας, αλλά στο περιεχόμενο. Η Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη μας υποσχέθηκε ότι θα αποτιμήσει την εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Ελπίζουμε να καταλήξουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι διακυβερνητικές συμφωνίες είναι λιγότερο αποτελεσματικές από την ε, κατάληξη και την ε, εφαρμογή κειμένων που έχουν συμφωνηθεί με την κοινωτική διαδικασία, δηλαδή με την συναπόφαση. Γιατί αυτή η διαδικασία επιτρέπει να υπάρχουν και οι σωστοί μηχανισμοί για να εφαρμοστούν οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι νομοθέτες που συμπεριλαμβάνουν και τα κράτη-μέλη και να υπάρχει σωστή λογοδοσία γιατί αν δεν υπάρχει σωστή λογοδοσία δεν υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών μας αυτή ήταν η πείρα μας από τα τελευταία χρόνια Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του για την αναθεώρηση τη οικονομική διακυβέρνηση και του πλαισίου τη και τι προκλήσει, τη λεγόμενη έκθεση Μπερέζ που εγκρίναμε τον παρελθόντα Ιούνιο, καλεί για ενισχυμένη δημοκρατική λογοδοσία μέσω μηχανισμών και σε ενωσιακό και σε κρατικό επίπεδο και για την πλήρη ένταξη του Δημοσιονομικού Συμφώνου στο ενωσιακό πλαίσιο. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, προσπαθεί να εγκαταλείψουν τα κράτη-μέλη την κυριαρχία τους. Είναι μια προσπάθεια να εφαρμοστούν οι βέλτιστοι κανόνες για να υπάρχει έλεγχος και διακυβέρνηση σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Πρέπει όλοι λοιπόν να κάνουμε περισσότερα, αλλά για να λειτουργήσει η Ευρώπη πρέπει ο δημοκρατικός έλεγχος και η επίβλεψη από τα κοινοβούλια να λειτουργεί αποτελεσματικά. Δεν θα δεχθούμε περισσότερη Ευρώπη, αν έχει ως τίμημα λιγότερη δημοκρατία, δημοκρατία λιγότερο κοινοβουλευτισμό. Αυτό θα ήταν συνταγή αποτυχίας. Η εμβάθυνση της ε, προσπάθειας συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής μπορεί να γίνει μόνο με τη στενή συνεργασία των εκλεγμένων εκπροσώπων των Ευρωπαίων πολιτών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε δημοκρατική λογοδοσία σε κάθε βήμα της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών προϋπολογισμών. Ως εταίροι σε αυτή την κοινή προσπάθεια για να τηρήσουμε τις αρχές του δημοκρατικού ελέγχου από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει λοιπόν όλοι, θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να κάνουμε περισσότερα για να λογοδοτεί ενώπιόν μα η εκτελεστική εξουσία. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε για αυτό τον κοινό στόχο. Επίση, Θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στη συζητήσεις σας σήμερα και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τη θαυμάσια συνεργασία και για τη θαυμάσια εργασία που επιτελέσαμε χθε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να δώσω το λόγο στην ε, συνάδελφό μου κυρία Αρίμπ. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρου του Ολλανδικού Κοινοβουλίου σας καλωσορίζω σε αυτήν τη διάσκεψη για την σταθερότητα, τον οικονομικό συντονισμό και την διακυβέρνηση που για μεγαλύτερη ευκολία ονομάζουμε διάσκεψη για το άρθρο 13. Εισαγωγικά λοιπόν τα σχόλιά μου. Οι πέντε άλλες κοινοβουλευτικές διασκέψεις που οργανώνει το Ολλανδικό Κοινοβούλιο θα λάβουν χώρα στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο όπου η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεδριάζουν στην καρδιά λοιπόν της Ολλανδικής Δημοκρατίας. Εδώ και μερικά χρόνια όμως η διάσκεψη για το άρθρο 13 γίνεται το πρώτο εξάμεινο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για αυτό. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία που μας οδηγεί σε αυτή τη διάσκεψη. Κάτω χώρες έχουν αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο της ιστορίας μας όπου οι χώρες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν μόνες τους. Πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα οι επιθέσεις στο Παρίσι, το προσφυγικό, είναι πράγματα που καταδεικνύουν κατάφορα αυτή την κατάσταση και είναι και τα πιο δύσκολα. Το θέμα της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δημοψήφισμα στις κάτω χώρες όσον αφορά την εταιρική μας σχέση με την Ουκρανία, είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στους πολίτες, περισσότερο από ποτέ. Και είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί μια χώρα να διαχειριστεί μόνη της. Χρειάζεται λοιπόν ευρωπαϊκή συνεργασία. Πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι και το θέμα της κοινοβουλευτικής διάσκεψης της Ολλανδικής Προεδρίας. Δηλαδή μαζί να οικοδομήσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κοινοβούλια έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο οι εθνικοί αντιπρόσωποι είναι σε καλύτερη θέση να γεφυρώσουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους πολίτες και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν ελέγχουν μόνο τη δικιά τους κυβέρνηση, αλλά μπορούν επίσης να φροντίσουν να σακωστεί η φωνή των πολιτών τους και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έμεσα ή Σήμερα θα συζητήσουμε για την οικονομική διακυβέρνηση και τη δημοσιονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το θέμα δηλαδή πάνω στο οποίο οργανώθηκε η συνεργασία μας ήδη από το 1952 με τη συνθήκη Ανθρακά και Χάλιβα. Σίγουρα είναι και δεολογικό θέμα, αλλά κυρίως είναι οικονομικό. Η διάσκεψη αυτή για το άρθρο 13 μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως τεχνική. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συζήτηση που θα έχουμε σήμερα έχει να κάνει με την ίδια την ευημερία μας. Θέλουμε δηλαδή υγιή και σταθερά δημοσιονομικά. Τα τελευταία χρόνια δουλέψαμε σκληρά γι' αυτό. Δεν ήταν εύκολο. Μερικές φορές είχαμε την εντύπωση ότι πηγαίναμε αντίθετα στο ρεύμα προκειμένου να τιμήσουμε τις συμφωνίες για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έχουμε δεσμευτεί νωρίτερα να τηρήσουμε είτε από το 1997 το σύμφωνο αυτό και να φροντίσουμε να βάλουμε το χρέος υπόελεγχο. Μερικές φορές ήταν δύσκολο να επικοινωνήσουμε όσον αφορά την ανάγκη για οικονομίες και ακόμα υπάρχουν δυσκολίες σε μερικές χώρες. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, καταφέραμε να πετύχουμε ευρεία συνένεση. Μέσα στον ΟΣΑ ε, μεταξύ άλλων φάνηκε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Το πετύχαμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Μετά από πολλές συζητήσεις για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική και δημοσιονομική κρίση, πλέον η προτερότητα βρίσκεται στο τι θα κάνουμε μακροπρόθεσμα. Φυσικά, η Ευρώπη είναι εδώ και τώρα και πρέπει να δράσουμε τη στιγμή που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα. Συγχρόνως όμως είναι δικιά μας ευθύνη, ναι, δικιά μας ευθύνη, επιμένω, ημών Ευρωβουλευτών, να σχεδιάσουμε το μέλλον. Αυτό μπορεί να ακούγεται πιο αφαιρημένο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Σε συνεργασία λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσαμε στην πράξη να δώσουμε ουσία στη διάσκεψη αυτή. Γι' αυτό και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε συζήτηση για τις επενδύσεις. Επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάπτυξη, θα συζητήσουμε για την ανταγωνιστικότητα επίσης και η συζήτηση αυτή θα γίνει κάπως διαφορετικά από ό,τι συνηθίζαμε μέχρι τώρα. Επίσης θα συζητήσετε και για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Ένα θέμα πολύ σημαντικό. Στα πλαίσια αυτά είναι το εξή. Υπάρχει αρκετός χώρος για την διακοινοβουλευτική συνεργασία και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στις κάτω χώρες έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Γιατί είμαστε χώρα μετά από δύσκολα μέτρα μπόρεσε να οικοδομήσει μια καλή παράδοση ισορροπίας με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Οικονομικού Σχεδιασμού που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για μας. Τέλος στη συζήτηση θα συμπεριληφθεί και η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Πώς εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις στις διάφορες χώρες μέλη. Πώς γίνεται ο δημοσιονομικός συντονισμός, μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο χωρίς να διαβρωθεί ο κοινοβουλευτικός ε, έλεγχος. Όλες αυτές είναι πολύ βασικές ερωτήσεις που πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί. Θα γίνει η συζήτηση λοιπόν έτσι όπως αντιστοιχεί σε μια αντιπροσωπευτική και σύγχρονη δημοκρατία με διαφάνεια. Θα δοθεί χώρος την διάδραση. Θα έχουμε, ελπίζω, επικοδομητική συζήτηση ποιότητας. Σας εύχομαι λοιπόν μια καλή συζήτηση που να επικεντρωθεί στον ορίζοντα που έχουμε μπροστά μας και που θα βασιστεί στην ιδέα ότι η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο ή τέλος πάντων πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ότι το σύνολο των χωρών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Gualtieri äh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφε. Να σας δώσω μια πληροφορία με ενημερώνουν ότι φέτος έχουμε 137 βουλευτές παρόντες. Ε, πρόκειται για αριθμό ρεκόρ. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσία σας ε, και για την ε, αντοχή σας που αντέχετε να μείνετε μέχρι τέλους εδώ στην αίθουσα. Βάσει διαδικασίας τώρα θα συνεχίσουμε με δύο συμπροέδρους, τον κύριο Μπάκερ, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Ολλανδικής Γερουσίας και του κύριου Ρομπέρτο Γκαλτιέρη, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους οποίους καλώ να έρθουν εδώ στο βήμα. Thank you, Mr. Schultz. Ευχαριστούμε τον κύριο Σούλτ και την κυρία Ρίπ ε, για τις αγωγές τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, τη συνεδρίασή μας. Αναμφίβολα οι απόψεις του κυρίου Σόουλτς και της κυρίας Αρίτ ε, θα βαρύνουν τις σημερινές συζητήσεις και βεβαίως ε, χαιρόμαστε που μας φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ στο ημικύκλιο. Βλέπω και κάποια μέλη του Κοινοβουλίου που ήταν παρόντα και χθε και φυσικά θα μας ε, φέρτε και την εμπειρία από τις χθεσινές συνεδρίες. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο πρώτο τμήμα στις βέλτιστες πρακτικές και ε, θα ήθελα να συμμετέχετε ενεργά και στις σημερινές συζητήσεις. Φαντάζομαι ότι έχετε λάβει το επεξηγυμνατικό σημείωμα που δόθηκε πριν από τη συνεδρίαση και περιμένω το έχετε διαβάσει κιόλα. Αλλά για όσους δεν είχαν αρκετό χρόνο να το διαβάσουν, θα συνοψίσω και θα σας πω ότι φύγει κάποια ζητήματα. Ποια είναι η παρούσα εμπειρία μας, ε, πώς ε, σχετίζονται τα κριτήρια μεταξύ τους στην πράξη και πώς ε, αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη κόστος όπως την αύξηση του κόστους για τα συστήματα υγείας και τα συντάξεις και κατά πόσον παρέχεται αρκετό περιθώριο για τις διακοινοβουλευτικές πρακτικές και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ε, τις ε, συστάσεις του Συμβουλίου και το πώς μπορούμε να τις κάνουμε κτήμα μας σε πολιτικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. είναι η καλύτερη μέρα για να σχεδιάσουμε αυτή τη συνεδρίαση, διότι στις 11 Φεβρουαρίου είχαμε τη συνεδρίαση του Eurogroup και δεδομένου ότι έχουμε εδώ τον κύριο Ντάισελ Bloom θα μάθουμε από πρώτο χέρι τι συνέβη σε αυτή τη συνεδρίαση, διότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα όσα ε, υπόθησαν ε, ε, πριν από σήμερα. Έχουμε επίσης και τον κύριο Κέις Βέντριγκ, ο οποίος είναι από το Ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο και θα μας πει για τον μηχανισμό εποπτείας. Επίσης, να καλωσορίσω την κυρία Βαλερή Ραμπό, Γενική Συγγήτρια της Επιτροπής Οικονομικών της Γαλλικής Εθνικής Συνέλευσης. Συγγνώμη που σας καλωσορίζω στα αγγλικά και θα μας εξηγήσει πώς αντιμετωπίζει η Γαλλία τις πρόσφατες οικονομικές προκλήσεις ε, σε σχέση με τα θέματα που συζητούμε σήμερα. Και τέλος, ε, να καλωσορίσω και τον συμπρόεδρό μου, το, ο οποίος με καλωσορίζει και αυτό σε μένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένω είναι εδώ με διπλή ιδιότητα, διότι θα κάνει και μία παρέμβαση επί του ουσίας. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο στους ε, ομιλητές μας, να σας πω δύο λόγια για το στόχο της σημερινής συνεδρίασης και να συνεισφέρω και εγώ το λιθαράκι μου. Οι διοργανωτές και εγώ συμμετείχα στην Οργανωτική Επιτροπή θεώρησαν ότι ε, και η ώρα να ανταλλάξουμε ε, πρακτικές εμπειρίες ε, μετά από κάποια χρόνια πλέον ενασχόλησης με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο για κάποιους από εμά το γεγονός ότι ζούμε σε καιρούς ε, υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και μάλιστα ε, και εντός των καθορισμένων δικτών του Δημοσιονομικού Συμφώνου σημαίνει ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε πλέον τις εμπειρίες μας. Θα σας πω και εγώ λοιπόν ε, σύντομα κάποιες από τις προσωπικές μου εμπειρίες και αυτή θα είναι και η μόνη παρέμβαση επί της ουσίας που θα κάνω. Ως ε, υπεύθυνο ε, επιπροπολογισμού στην Ολλανδική Γερουσία γιατί ε, ο κόμμα μου, εμείς έχουμε ένα σύστημα δύο βουλών στην Ολλανδία. Οι δύο πρόεδροι των, της, τα δύο όργανα έχουν και τα δύο δυνατότητα νομοθετικών προτάσεων και κάθε πρόταση που υποβάλλεται θα πρέπει να περάσει με πλειοψηφία και από τις δύο βουλές. Στην πρώτη χρονιά που ανέλαβα τον προπολογισμό, είχα μια αίσθηση εξωτερικής παρέμβασης. Ε, επειδή υπήρχε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προβλέψιμο κύκλο προπολογισμού. και μάλιστα υπήρχαν και κάποιες πιέσει. Υπήρχε μια παρέμβαση με τις ε, συστάσεις ε, αναχώρα, οι οποίες θα έπρεπε να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες προτάσεις στον προπολογισμό και το κατά πόσο θα υπάρξει συμφωνία ή όχι. Και στην αρχή, ε, στον πρώτο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ολλανδική Κυβέρνηση, και νομίζω ότι μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Υπουργό Οικονομικών αυτών, ε, δεν υπήρχε μια ασφαλή πλειοψηφία και στις δύο βουλές ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές για πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το συνταξιοδοτικό. Ε, στεγαστικά δάνεια, ηλικίες ταξιοδότησης, ε, για να σας αναφέρω μερικά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο αποδείχθηκε ότι έχει και πλεονεκτήματα αλλά και κάποιες αδυναμίες. Πλεονεκτήματα είναι, ε, θα έλεγα, το γεγονός ότι η συνθήκη έχει ε, προσθέσει μια εξωτερική ε, πειθαρχία, ένα εξωτερικό σημείο αναφορά το οποίο βασίζεται σε εξωτερική ανάλυση που σημαίνει ότι λαμβάνονται μέτρα που ορισμένες φορές είχαν καθυστερήσει ήδη ε, πολύ. Η αδυναμία του είναι ακριβώς το ίδιο σημείο και οι περισσότεροι θα το έχετε βιώσει. Η αδυναμία είναι ότι υπάρχει ορολογία με την οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι, νέες παρεμβάσεις ε, στο σημερινό κύκλο. Ε, υπάρχει υλικό ε, βιβλιογραφία και μια ε, πολιτική επιλογή αυτή τη στιγμή για λιτότητα. Εγώ ειλικρινά συμφωνώ με αυτή την επιλογή, αλλά συνειδητοποιώ επίσης ότι αυτό βρίσκεται κέντρο της πολιτικής συζήτησης σε κάθε χώρα. Και φυσικά ο καθής μπορεί να εξοικειωθεί και με την ορολογία και με το κύκλο ε, προϋπολογισμού και το έλλειμμα, αλλά κάποια πράγματα είναι πράγματα με τα οποία δεν έχουμε εξοικειωθεί ακόμα. Και εδώ έχουμε ένα από τα θέματα που θα κάνουμε στη σημερινή συζήτηση. Η νομιμοποίηση των ε, μακρόπνων συνεπειών του κύκλου αυτού. Και πιστεύω ότι ε, εμείς εδώ με αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο, διότι στην ουσία πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία ε, της αδιάφανης διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η απουσία άλλων δημοκρατικών ε, θεσμών αποδυναμώνουν την νομιμοποίηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Επομένως, τα θέματα τα οποία μας ε, αφορούν στον κύκλο προπολογισμού είναι πάρα πολύ σημαντικά και σε εθνικές πολιτικές συζητήσεις. Πολλοί από εσά, κυρίω από χώρε που έχουν λάβει δραματικά μέτρα, ε, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη θα έχουν σίγουρα πράγματα να συνεισφέρουν και να μας πούν σήμερα. Και σήμερα βρισκόμαστε στο κατάλληλο βήμα και έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά μεταξύ μας και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιλήψουμε και διδάγματα ο ένας από τον άλλον σήμερα και αυτός είναι και ο στόχος της πρωινής συνεδρίασης. Να περάσω τώρα σε κάποια πρακτικά ζητήματα. Θα γνωρίζετε πώς μπορείτε να λάβετε το λόγο. Αφού ε, μιλήσουν οι τέσσερις ομιλητές, ε, θα φροντίσουμε να μιλήσουν όσο το δυνατόν ε, περισσότερα μέλη. Αλλά φυσικά υπάρχει και χρονικός περιορισμός και πρέπει να διαχειριστούμε καλά το χρόνο μου. γι' αυτό σας ζητώ να μας βοηθήσετε κι εσείς να τηρήσουμε τα χρονικά όρια όταν χρειαστεί. Δύο ή τρία λεπτά ανάλογα με τον αριθμό των ομιλητών και θα είμαστε αυστηροί, όσο το δυνατόν πιο αυστηροί. Έχετε όλοι ε, το έντυπο για να μιλήσετε, επομένως συμπληρώνετε το έντυπο και μας κοινοποιείτε την επιθυμία σας να λάβετε το λόγο. Και αυτό ισχύει και για τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και φυσικά και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας φιλοξενεί. δύο εθνικοί βουλευτές ε, και ακολουθεί ένας ευρωβουλευτής. Αν χρειαστεί να προσαρμόσουμε βέβαια τον τύπο θα τον προσαρμόσουμε, αλλά έτσι θα ξεκινήσουμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γέρουν Ντάισελμπλουμ, ε, τον προειδοποιώ όμω θα είμαι αυστηρό με το χρόνο για τα 10 λεπτά, όπω είναι και ο ίδιο με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μπορώ κάπου να βλέπω το χρόνο που μου μένει. Θα σας υπενθυμίσω, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας σε αυτήν την διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη. Πολύ χρήσιμο βήμα. Από πλευρά της Ευρωζώνης μπορούμε μόνο να ωφεληθούμε από τη στενή συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων του λαού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και διαμορφωτών της πολιτικής. Πρώτα απ' όλα να σας παρουσιάσω την οικονομική κατάσταση. Ως Υπουργός Οικονομικών που με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πάντα θέλω να αναφέρομαι στην οικονομική κατάσταση πριν ασχοληθώ με την έκθεση των πέντε προέδρων και την εργασία που πρέπει να κάνουμε για την οικονομική διακυβέρνηση. Η Ευρωζώνη κατάφερε να υπερβεί την κρίση στα χρηματοπιστωτικά και του δημοσίου χρέους χάρη στην αποφασιστική εφαρμογή πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Μαζί με καινοτόμε ε, προσπάθειες από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για να προστατεύσουν το ενιαίο νόμισμα. Είμαστε τώρα την τρίτη χρονιά ανάκαμψη ως Ευρωζώνη και διευρύνεται αυτή η ανάκαμψη σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Αλλά αυτή η ανάκαμψη ε, εξαρτάται ακόμη πολύ από διάφορε αναταράξεις. Χαμηλέ τιμέ πετρελαίου, ε, πολύ γενναιόδορη νομισματική πολιτική για την, ε, για την ισοτιμία μας. Επίσης έχουμε και εξωτερικές απειλές όπως η επιβράδυνση στην Κίνα και διάφοροι τριγμοί σε άλλε εξωτερικέ αγορέ. Άρα πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη για να γίνει ανατροφοδοτούμενη η ανάκαμψη. Έχουμε ακόμη πολλά μεγάλα, σε πολλέ χώρε υψηλά ποσοστά ανεργία και προβλήματα με την οικονομική απόδοση πολλών περιοχών τη Ευρωζώνη. Άρα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εφησυχασμού. Οι, πρόσφατε οι πρόσφατες ε, στα χρηματιστήρια αποδεικνύουν ότι σε πολλούς τομείς πρέπει να κάνουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσουμε τους κανόνες της Τραπεζικής Ένωσης. Ω πρόεδρος του Eurogroup και του ECOFIN υποστηρίζω πλήρω, πρωτοβουλία τη Κομισιόν για να δημιουργηθεί ε, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, ούτως ώστε να υπάρξει περισσότερη δυνατότητα χρηματοδότησης τη πραγματική οικονομία και για να ενισχύσουμε την Τραπεζική Ένωση για να αυξηθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και να σταματήσει ε, αυτός ο φαύλος κύκλος των κρίσεων δημοσίου χρέους. Η ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης δεν σημαίνει μόνο ότι θα έχουμε ένα σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων και ένα ταμείο εξυγείας των τραπεζών, αλλά επίσης αποφασιστική πρόοδος για τη μείωση των κινδύνων και πιο ισορροπημένες συνθήκες ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες. Οι κίνδυνοι θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπιστούν εκεί που προκύπτουν. Ένα στόχο τη Τραπεζική Ένωση είναι να μην χρειαστεί να διασώσουν ε, χρεοκοπημένε τράπεζε στο μέλλον ή φορολογούμενοι. Και η οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών είναι ένα καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η συνέχιση της σύγκληση είναι βασικό θέμα της έκθεση των πέντε προέδρων. Η έκθεση έχει τίτλο «Ολοκλήρωση της ε, ΟΝΕ» και είμαι ένας από του συντάκτε με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των άλλων θεσμικών οργάνων. Στόχο τη ε, έκθεση αυτή είναι να υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ ρεαλισμού και μακρόπνοου οράματο, που να έχει μια σταδιακή προσέγγιση. Για το πρώτο στάδιο μέχρι τα μέσα του 2017 προτείνει διάφορα βράχυπρόθεσμα μέτρα, ούτω ώστε η Ευρωζώνη να γίνει πιο ανθεκτική με ένα σωστό νομικό πλαίσιο. Θέλουμε δηλαδή να διορθώσουμε δημοσιονομικούς, δημοσιονομικές ε, και ε, φορολογικές ανισορροπίες. Και θέλουμε επίσης οι ευρωπαϊκές ε, συστάσεις πολιτικής να γίνονται πιο αποδεκτές από τα κράτη-μέλη και να υπάρχει δημοκρατική λογοδοσία. Όλες αυτές οι πλευρές συνδέονται. Χρειάζεται λοιπόν παράλληλη πρόοδο σε όλους αυτούς τους τομείς για να διευκολύνουμε το πέρασμα στη δεύτερη φάση που θα έχει πιο μακρόπνοα μέτρα για να ολοκληρώσουμε την δομή της ΟΝΕ μέχρι το 2025 αυτή η διαδικασία. Θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα αλλαγέ στι συνθήκε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι το αργότερο μέχρι το τέλο του 2017 θα περάσει στην εξέταση των μέτρων για δεύτερη φάση. Και προτάσει τη Κομισιόν, ιδιαίτερα του Επιτρόπου Ντομπρόφσκη για το πρώτο στάδιο, μέχρι στιγμή δεν έχουν βρει ευρύ ανταπόκριση. Το Eurogroup και το Συμβούλιο Κοφίν και διάφορα προπαρασκευαστικά σώματα εξετάζουν προσεκτικά τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να εφαρμόσουν τις προτάσεις για το πρώτο στάδιο. Μία από αυτές τις προτάσεις είναι η δημιουργία εθνικών επιτροπών ανταγωνιστικότητας. Οι αρχές ανταγωνιστικότητας, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καθορίζουν με, σωστούς, με σωστές παραμέτρους την εθνική συζήτηση, ούτως ώστε να διευκολύνουν τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια να καταλήγουν στις σωστές αποφάσεις. Αυτή, αυτές οι επιτροπές ανταγωνισμού μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια μεταρρυθμίσεων, κυρίω σε εθνικό επίπεδο. Να βελτιώσουν το σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι σημείο κλειδί. Πώ θα βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα του κοινωνικού μα προτύπου. Πώ θα βελτιώσουμε την απασχολησιμότητα. Διασφαλίζοντα όμω ότι έχουμε ένα σωστό προπολογισμό. Αυτέ οι εθνικέ επιτροπέ δεν θα είναι κίνδυνο για τι συλλογικέ διαπραγματεύσεις γιατί αυτός ο κίνδυνος ε, αναφέρθηκε, θα είναι για να ενισχύσουν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και ενισχύουν την εσωτερική ζήτηση. Και χρειάζεται και ανεξάρτητη δυνατότητα παροχής συμβουλών και επίσης ανταλλαγή πρακτικών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα δίκτυο εθνικών επιτροπών ανταγωνιστικότητας για όλη την Ευρωζώνη. Τώρα να στραφώ στον ζωτικό ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων για την οικονομική διακυβέρνηση. Για να είναι αποτελεσματικά τα μέσα μας και για να επιτύχουμε στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής ΟΝΕ είναι θεμελιώδες να συμμετάσχουν τα εθνικά κοινοβούλια. Διότι, σε τελευταία ανάλυση, τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ οικονομικές προκλήσεις πρέπει να βρουν στήριξη και να εφαρμοστούν από τα εθνικά κοινοβούλια. Από φέτος και στο εξή θα προσπαθήσουμε να περιλαμβάνουμε στο πλαίσιο οικονομικού συντονισμού μέσω συστάσεων προ την Ευρωζώνη όλα αυτά τα στοιχεία στην αρχή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Με αυτόν τον τρόπο οι συστάσει για την Ευρωζώνη μπορούν κατόπιν να ενταχθούν στι ε, ειδικέ αναχώρα συστάσει, οι οποίε ε, εκδίδονται τον Μάιο. Οι συστάσει για την Ευρωζώνη ε, καλούν επίση για να υπάρξει περισσότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μέσω ανταλλαγή εμπειριών από χώρα σε χώρα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και για να υπάρχει περισσότερη έμφαση στην, ε, στον καθορισμό προτύπων από χώρα σε χώρα. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τιμών αναφοράς. Γι' αυτό η συζήτηση για την, ε, τον σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων συζητώνται συχνά στο Eurogroup. Τα τελευταία χρόνια σημειώσαμε πρόοδο στον τρόπο συντονισμού των οικονομικών μας πολιτικών. Αλλά μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για την εφαρμογή των οικονομικών αυτών πολιτικών η εφαρμογή των αναχώρα συστάσεων μπορεί να βελτιωθεί. Πρώτα απ' όλα περιορίζοντας τον αριθμό των συστάσεων. Αν δείτε πόσες συστάσεις ε, εκδίδονται από τα διάφορα κράτη-μέλη, θα καταλάβετε τι εννοώ. Δεύτερον, πρέπει να είναι πιο στοχευμένες στα ζωτικά στοιχεία. Αυτά που πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα αναχώρα. Επίσης απαιτείται περισσότερη εθνική αποδοχή. Πολλά κράτη-μέλη απλώ σημειώνουν τι συστάσει αυτές, τι λαμβάνουν υπόψη και συνεχίζουν τα εθνικά τους προγράμματα και τις εθνικές τους προτεραιότητε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Τρίτον, η αναχώραση στάσης δεν θα πρέπει να είναι σε αιτήσια βάση. Θα μπορούσε να εκδίδονται σε πολιετή βάση. Γιατί όπω ξέρετε, οι κυβερνήσει συνήθω ε, έχουν θητείε τριών, τεσσάρων, πέντε ετών. Ούτω ώστε να έχουν χρόνο οι κυβερνήσει να εφαρμόσουν ένα σύνολο συστάσεων που έχουν συζητηθεί με την Επιτροπή, με τα κοινοβούλια και τα εθνικά και το δικό μα εδώ. Το δικό σα εδώ. Ο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων για να δημιουργηθεί αυτή η εθνική αποδοχή είναι απαραίτητο. Αλλά πρέπει να συμμετάσχουν και οι κοινωνικοί εταίροι. Τώρα, το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρω τι ε, αρμοδιότητε που προβλέπονται από τη συνθήκη για την δευτερογενή νομοθεσία, ιδιαίτερα στα πλαίσια του οικονομικού διαλόγου. Το Κοινοβούλιο ήδη δρά με αυτόν τον τρόπο και με το πνεύμα τη έκθεση των πέντε Προέδρων το πράττει όλο και περισσότερο. Πρόσφατα συζήτησε τι ε, προτάσει ε, για την Ευρωζώνη τη Κομισιόν για το 2016 και είχα το προνόμιο να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση στην Ολομέλεια μαζί με τον ε, πρόεδρο Γιούγκερ και τον αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάντα αποδέχομαι τέτοιε προσκλήσει όπω και τι προσκλήσει τη Επιτροπή Οικονομικών του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτόν τον τρόπο έχουμε ήδη αρχίσει να εφαρμόσουμε, να εφαρμόζουμε την έκθεση των πέντε πρόεδρων που καλούν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και του Συμβουλίου να συμμετέχουν δια διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Για να έχουμε λοιπόν καλύτερο διάλογο. Ανέλαβα την πρωτοβουλία να αυξηθεί η διαφάνεια και των ε, συνεδριάσεων του Eurogroup. Κύριε Πρόεδρε, εσεί αναφερθήκατε στον διαφανή τρόπο λειτουργία του Eurogroup. Από εδώ και το εξή, πριν από τι συνεδριάσει μα, θα δημοσιεύουμε πιο αναλυτική και σχολιασμένη ημερήσια διάταξη και θα δημοσιεύουμε επίση λίγο μετά τι συνεδριάσει μία συνόψηση των πορισμάτων μας. Επίσης θα πιέσουμε ούτω ώστε να δημοσιοποιείται ταχύτατα οποιοδήποτε έγγραφο συζητούμε στη συνεδριά μας. Όλα αυτά θα κάνουμε φυσικά σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα που μας παρέχουν αυτά τα έγγραφα. Ως Eurogroup και πρόεδρος, ως πρόεδρος του Eurogroup και του ECOFIN θα κάνω κάθε προσπάθεια να διευρυνθεί η συζήτηση, να διευκολυνθούν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν ούτως ώστε να υπάρξει εθνική αποδοχή των προγραμμάτων να υπάρξει ευαισθητοποίηση για να ενισχυθεί η ε, πολιτική και δημόσια αποδοχή των προσπαθειών μεταρρυθμίσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι και προς το συμφέρον των κρατών μελών και προς το συλλογικό μας συμφέρον και ελπίζω η σημερινή σας συνεδρίαση να είναι χώρος όπου θα προκύψουν πολλές νέες απόψεις για τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Ντάσερμπλουμ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Κέις Φεντρίκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, καλημέρα. Σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θα μιλάω γρήγορα, λέει ο μιλητή. Κυρίε και κύριοι. Αλλά όχι πολύ γρήγορα, εντάξει. Όχι. Κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από θεμελιώδεις αλλαγές ήδη από τη δεκαετία του 90. Από τότε που ξεκίνησε η οικονομική και δημοσιονομική κρίση το φθινόπωρο του 2008, η ΟΝΕ βρέθηκε υποπίεση, όπως όλοι γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε την ΟΝΕ και την Ευρωζώνη και πάλι και προσπαθήσαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για να ανταποκριθούμε λοιπόν σε αυτή την κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Ευρωζώνης ξεκίνησαν με νέες πολιτικές και μεταρρυθμιστικές ε, πολιτικές. Νέες πολιτικές λοιπόν με διαβουλεύσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ώστε να στηριχτούν κάποιες χώρες. Υπήρξε νέο ταμείο για να στηρίξει τις τράπεζες της Ευρωζώνης και όλα αυτά από την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι, οι δημοσιονομικοί κανόνες εισήχθησαν προκειμένου να ενισχυθεί η νομισματική ένωση. Δημοσιονομική εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης των χωρών μελών και μακροοικονομική επίβλεψη των χωρών μελών. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το Σεπτέμβριο του 2014 το ελεγκτικό συνέδριο των κάτω χωρών ετοίμασε έκθεση με νέους δημοσιονομικούς και οικονομικούς κανόνες προκειμένου να ενισχυθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Το ζήτησε το Γερουσία και υπήρχαν συνέπειες και στις κατοχώρες αλλά και σε όλες τις χώρες μέλη. Οι κανόνες αυτοί όμως κυρίως έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και γι' αυτό αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε μια ευρύτερη προσέγγιση που να συμπεριλαμβάνει και τις χώρες μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για την ε, συμμόρφωση λοιπόν θελήσαμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και να πάρουμε μαθήματα για το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν κάποια από αυτά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε να μοιραστώ μαζί σας. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα της έρευνά μας. Κάποια από αυτά έχουν πρόσφατα επικαιροποιηθεί. Εδώ όπως βλέπετε πρόκειται για ένα πυκνά αποτελέσματα. Βλέπει εδώ πότε χώρες μέλη βρέθηκαν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Το βλέπετε αυτό σε κίτρινο. Και τότε το Συμβούλιο έπρεπε να πάρει μέτρα. Αυτό το βλέπετε σε πορτοκαλί. Έτσι λοιπόν υπήρχε επίβλεψη που δεν υπήρχε στην αρχή από τις ε, χώρες ε, μέλη όλες. Οι οικονομικές ε, κυρώσεις δεν είχαν επιβληθεί. Οι χώρες οι οποίες δεν ανταποκρινόντουσαν στις προδιαγραφές πήραν κάποια αναβολή. Αυτό όμως άλλαξε από τη στιγμή που εισήγαγαμε νέα μέτρα από το 2010. Πρόσφατα λοιπόν ο αριθμός των χωρών που βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος έχει μειωθεί. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ συχνά αποφάσισε να μην αρχίσει τη διαδικασία εξαιτία ειδικών συνθήκων που προσωρινά μείωναν την δημοσιονομική πειθαρχία. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι τα μέτρα αυτά που ενισχύουν τις μακροοικονομικές πολιτικές των χωρών μελών οδήγησαν σε ένα σύνολο περίπλοκων ρυθμίσεων και νομοθεσιών. Και ακριβώς αυτό το γεγονός ότι πρόκειται για πορύπλοκους κανόνες μας οδήγησε σε μεγαλύτερη δυσκολία εφαρμογής. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Είναι επίσης σαφές ότι εξαιτία αγωγή των νέων κανόνων, ε, τη συμφωνία τη της των 6 και των 2 ε, διών, όλες οι χώρε μέλη λογοδοτούν τώρα για τις μακροοικονομικές τους και δημοσιονομικές τους πολιτικές. Όμως η δυνατότητα de facto της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλάξει τις πολιτικές των χωρών μελών είναι κάτι περιορισμένο. Γιατί τελικά είναι οι χώρες μέλη εκείνες οι οποίες παίρνουν τις αποφάσεις. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια τώρα όσον αφορά τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πώς η νέα διαδικασία έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Η διαδικασία ήταν ε, περιορισμένη στα στάδια της πρόληψης με περιορισμένο αριθμό χωρών. Όμως οι χώρες με, υπερβολικό, με υπερβολικές ε, ανισορροπίες αυξήθηκαν από το 2014 στο 2015. Η διαδικασία πάντως δεν ενεργοποιήθηκε. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα σε κάθε στάδιο της ε, διαφορετικής διαδικασίας αποφασίζει για το πόσο σοβαρή είναι η ανισορροπία, ποια είναι η φύση της ανισορροπίας, αλλά τα κριτήρια δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λοιπόν συνεχίζουν να αναπτύσσουν τις δυνατότητε αυτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε συζήτηση για την εναρμόνιση του συστήματος αναφοράς των χωρών μιλών, ενισχύοντας τη λογοδοσία ώστε να υπάρξει καλύτερη συγκρισιμότητα μεταξύ των χωρών μελών στι δημοσιονομικέ του πολιτικές. Αυτό για μα είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το τελικό θέμα, το τελευταίο μου, είναι το εξής. Η καλή διακυβέρνηση, ο δημοκρατικός έλεγχος, η λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο παντού στο Eurogroup και στον ε, Πρόεδρο. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα, για την μακροοικονομική μας πολιτική. Κυρίες και κύριοι, όταν η έκθεσή μας πριν από ένα χρόνο ε, δημοσιεύτηκε, μας οδήγησε να πάρουμε κάποια μαθήματα για το μέλλον. Και αυτό θα πω και τώρα σε εσά. Διαπιστώνουμε ότι οι χώρες μέλη δεν συμμορφώθηκαν ικανοποιητικά με τους κανόνες που είχαν ε, προβλεφθεί ήδη πριν από το 2008. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αναγκάστηκαν να τους επιβάλλουν. Πρόκειται για περίπλοκους κανόνες, είναι αλήθεια, και δεν επιβλήθηκαν όπως θα έπρεπε τόσο αποτελεσματικά όσο χρειαζόταν για μια οικονομική διακυβέρνηση. Ο τελικός στόχος είναι η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης με εμπιστοσύνη των αγορών, του δημοσίου, των επιχειρήσεων, εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα εκείνη της Ευρωζώνης. Οι κανόνες, οι διαδικασίες απαιτούν πάνω απ' όλα διαφάνεια και απλοποίηση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Ο έλεγχος των ε, κοινοβουλίων πρέπει να γίνεται πιο ουσιαστικά με απλοποιημένες διαδικασίες όταν αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον, πολλά βήματα μπορούν να ληφθούν για την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία μικροοικονομικών ανισορροπιών. Το βαθμολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρινίζει τη σχέση των προσπαθειών που κάνουν οι χώρες μέλη με τα αποτελέσματα. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται διαφάνεια για το κοινό και για το κοινοβούλιο και θα ενισχυθεί αν δεν βασιζόμαστε μόνο στην οικονομική απόδοση αλλά και σε άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα όπως επίσης και με την εφαρμογή από τις χώρες μέλη των ε, ειδικών αναχώρας συστάσεων. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση δίνει όλο και περισσότερη σημασία στα υγιή δημοσιονομικά. Οι διαστροτικές ε, ανισορροπίες παρατηρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό μίλησα πριν για εναρμόνιση των ε, κανόνων αναφοράς των ε, στοιχείων που αφορούν την κάθε χώρα. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους βουλευτές και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για σας να μπορέσετε να καταλάβετε περισσότερο με διαφάνεια τις αλλαγές στα δημοσιονομικά. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Περισσότερη και βουλευτική προσοχή λοιπόν για αυτό το ζήτημα των ανισορροπιών. Τέλος θέλω εδώ να πω ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην ε, διακυβέρνηση του Eurogroup και στην διαφάνεια όσον αφορά τη λειτουργία του. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος του Eurogroup, την διαφάνεια του Eurogroup την έχει βάλει στην ατζέντα της συνεδρίασης της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η Προεδρία του Eurogroup δεν έχει καθεντρηθεί απόλυτα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μέλλον θα αποφασιστεί κατά πόσο θα υπάρχει ένας μόνιμος πρόεδρος ή όχι. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κλείσω εδώ την παρουσίασή μου με ένα δίλημα. Προφανώς είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί ικανοποιητικά η Ευρωζώνη. Η οικονομία των χωρών αυτών, αλλά και το μέλλον των πολιτών της Ευρωζώνης εξαρτάται ακριβώς από αυτή την κατάσταση. Για να λειτουργήσει λοιπόν καλά η Ευρωζώνη χρειάζεται ενίσχυση της δημοσιονομικής ισορροπίας στις χώρες μέλη. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει απόλυτα σήμερα. Έχουμε δει κατά το παρελθόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την προσέγγιση λειτουργία βάση κανόνων από τι χώρε μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών εισάγοντας περισσότερου κανόνε ή κάνοντα πιο αυστηρού του ήδη υπάρχοντε κανόνε με το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, για παράδειγμα. Η συμμόρφωση όμω των χωρών μελών με του κανόνε αυτού δεν είναι βέλτιστη για να το πω έτσι ήπια. Πολλοί κανόνες δεν εφαρμόζονται. Οπότε, τίθεται το ερώτημα, αυτή η προσέγγιση λειτουργία βάσει κανόνων είναι ο καλύτερο τρόπο για να συντονίσουμε τι οικονομίε των χωρών μελών, ή για να το πω διαφορετικά. Οι χώρε μέλη θέλουν πραγματικά οι ευρωπαϊκές οικονομίες να διευθύνονται σε ένα βαθμό από τι Βρυξέλλε, ή η Ευρωζώνη είναι τόσο περίπλοκη που είναι δύσκολο να υπάρχουν βιώσιμοι κανόνε και συντονισμό. Αυτό λοιπόν το δίλημα με αυστηρούς κανόνες από τη μία αλλά μη πλήρη συμμόρφωση προς την άλλη δεν βοηθάει να βελτιώσουμε και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των οικονομικών αγορών στην λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται συζήτηση για τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και τι πρέπει να κάνουμε για να είναι σε καλή κατάσταση η ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή είναι η συζήτηση λοιπόν και εσείς όσο βουλευτές μπορείτε να συνεισφέρετε τα μάλα. Ίσως είναι πολύ νωρίς βέβαια για να δοθεί απάντηση στο δίλημα αυτό. Τώρα βρισκόμαστε μετά την κρίση και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση εξακολουθεί να αναπτύσσεται με νέες διαδικασίες. Με νέες θέσεις, με νέες σχέσεις. Όλες αυτές οι νέες διευθετήσεις πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για να ανακτηθεί εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση για τη συζήτηση. Προτείνετε περισσότερες ε, αρχές ή περισσότερους κανόνες. Εγώ απλώ έθεσα ένα ερώτημα, όπως κάνουν ε, τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, εντάξει, μια δοκιμή έκανα. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βαλερή Ραμπό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα σε αυτή τη σύντομη εισαγωγή να αναφερθώ σε τρία σημεία. Καταρχάς, ε, την εμπειρία ε, της καθοδήγησης των δημοσίων δαπανών που κάναμε στη Γαλλία. Δεύτερον, τη σχέση με τον οικονομικό κύκλο και πώς τα ευρωπαϊκά εργαλεία τα οποία ε, χρησιμοποιήθηκαν μας βοήθησαν να ε, καθοδηγήσουμε τη διαδικασία και τρίτον, εδώ να συμφωνήσω και απόλυτα με τον πρόεδρο του Eurogroup που έλεγε ότι πρέπει να ε, σχεδιάσουμε καταλήλως τις μεταρρυθμίσεις και πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτή την αρχή. Πρώτο σημείο να σας πω τι συνέβη στη Γαλλία. Προηγουμένως είδατε ένα διάγραμμα το σύμφωνο για τη Γαλλία και για κάποιες χώρες οι οποίες δεν είχαν σεβαστεί πλήρως το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης ε, μας οδήγησε να ε, διαπιστώσουμε ότι εδώ και 10 χρόνια είχε είχαν αυξηθεί οι δημόσιες διαπάνες ε, στη Γαλλία κατά 35 περίπου δις ετησίως που σημαίνει 3,2% ε, του ΑΕΠ κάθε χρόνο σε αξία. Ε, εδώ και 10 χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που μας ε, επιτρέπουν να φέρουμε και πάρκες τις δημόσιες δαπάνες στο 0,9% σε αξία, που σημαίνει ότι είναι λιγότερο ε, γρήγορη από την πρόοδο του ΑΕΠ μας και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό ορόσημο. Ε, έγινε με πολύ ε, στεναρά μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τη διαχείριση των δημοσίων δαπανών ώστε να σταματήσουμε αυτή την αύξηση των δημοσίων δαπανών. Αυτό είναι το πρώτο σημείο και αυτό μας επέτρεψε επίσης ε, να μειώσουμε το δημόσιο έλλειμμα το ονομαστικά έλλειμμα, το οποίο ήταν περίπου ε, κάτι παραπάνω από το 10% στην αιχμή της χρήσης και τώρα είμαστε στο 4,2% και στόχο έχουμε να φτάσουμε στο 3,8% εφέτος. Εντάξει, είχαμε λοιπόν μια δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών, μειώσαμε τις πιστώσεις που δίνονται στις διάφορες διοικήσεις. Ένα δεύτερο ερώτημα λοιπόν που ετέθη στη συνέχεια είναι πώς διαρθρώνεται αυτή η πολιτική με την μακροοικονομική συζήτηση, δηλαδή με την υποστήριξη στην ανάπτυξη, υποστήριξη στη ε, δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι αναπόσπαστο τμήμα των βασικών ε, προγραμμάτων του Ευρώπη 2020. Εδώ η συνθήκη ε, μας έδωσε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο να μπορέσουμε να ε, κατευθύνουμε το διαρθρωτικό έλλειμμα. Δηλαδή, να μπορέσουμε να πούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στον οικονομικό κύκλο και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να μειώσουμε το νομαστικό έλλειμμα χωρίς να ανακόψουμε την πορεία της ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό και ενδιαφέρον μέσο, αλλά πρέπει να αναγνωρίσω ενώπιον σας αγαπητοί συνάδελφοι ότι δεν είμαι βέβαιη ότι έχει γίνει απόλυτα κατανοητό. Και τουλάχιστον ε, εντός της ε, Γαλλικής Εθνικής Συνέλευσης, ε, δεν θα ήθελα εδώ να προσβάλλω τους συναδέλφους, αλλά το πολύ δέκα βουλευτές έχουν αντιληφθεί ποιες είναι οι δυνατότητες Τη χρήση αυτού του εργαλείου του διαρθρωτικού ελλείμματο. Βλέπω τον πρόεδρο του Eurogroup να χαμογελά. Νομίζω ότι είναι από αυτά τα ερωτήματα που έπρεπε να τεθούν. Αυτό λοιπόν το διαρθρωτικό έλλειμμα και το, η χρήση του δεν έχει γίνει κατάλληλα αντιληπτό και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να μας δώσει λίγο περισσότερα εργαλεία για να μας πει πού βρισκόμαστε στον κύκλο και για μια δεδομένη χώρα, αλλά και για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση εδώ. Δεύτερον, ε, πάντα για το διαστατικό έλλειμμα, όταν η δράση είναι λίγο πιο βίαιη, αν θέλετε, μειώνεται με το δημοσ... οι δημόσιες δαπάνες, αλλά κατά συνέπεια έχουμε και πολύ σημαντική μείωση των επενδύσεων. Η ανάκαμψη όμως και η επιστροφή στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνοδεύεται από την αύξηση των επενδύσεων. Και νομίζω ότι αυτό καταστράφηκε στον τρόπο με τον οποίο προσπαθήσαμε να μειώσουμε το δημόσιο έλλειμμα, ίσως γιατί ε, αυτό το εργαλείο του διαρθρωτικού ελλείμματος δεν έχει γίνει κατάλληλα αντιληπτό, δεν έχει τεκμηριωθεί καταλήλως και θα μπορούσα να πω δεν έχει και μετρηθεί καταλήλως. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο λάβαμε υπόψη μας στη Γαλλία είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και εδώ συμφωνώ απολύτως με τον πρόεδρο του Eurogroup είναι σημείο ε, ζωτική σημασία. Πρόκειται για ένα στάδιο κλειδί ώστε να μπορέσουμε και να ε, κατευθύνουμε τα δημόσια οικονομικά αλλά να υποστηρίξουμε και την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς οι πέντε στόχοι που βρίσκονται στο θεματολόγιο του Ευρώπη 2020 δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν καταλήλω ε, στο δικό μα το κοινοβούλιο, στην Εθνική μα Συνέλευση. Πρόκειται για πέντε στόχους που είναι πολύ ακριβείς, ε, πολύ αναλυτικοί και που κατά την άποψή μου μπορούν να δώσουν μια όθηση στην ανάπτυξη στι χώρε μας. Πρόκειται για πέντε στόχους, ε, τους αναφέρετε και εσείς κύριε που είπατε δεν θα πρέπει να γίνονται πολλέ συστάσει και νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ μαζί σας. Αυτοί οι πέντε στόχοι λοιπόν πρέπει να διαβιβαστούν καταλήλω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα υπόλοιπα κοινοβούλια και να πούνε τι απαντήσει δίνουμε εμεί σε αυτού του πέντε στόχου, τι απαντήσει μπορούμε να δώσουμε ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε στον οικονομικό κύκλο, διότι δεν βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο σημείο στη χώρα μα. Νομίζω ότι όλα αυτά, και με αυτό ολοκληρώνω, ε, αξίζουν να χρησιμοποιηθούν με πολύ πιο επιθετικό τρόπο ε, και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα εθνικά μας κοινοβούλια ώστε να μπορέσουμε να πούμε ποιες είναι οι δράσεις που θα υλοποιήσουμε προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους αυτού του θεματολογίου 2020 και πού θα περιοριστούμε, δηλαδή πού βρισκόμαστε στον οικονομικό κύκλο. Ε, θα ολοκληρώσω αυτό κύριε Πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι μας έχετε δώσει κάποια ουσιαστικά στοιχεία με αυτούς τους στόχους Ίσως ε, θα χρειαζόμασταν ε, λίγα περισσότερα κίνητρα, ένα ένασμα για να τα χρησιμοποιήσουμε με πιο αποτελεσματικό και επιθετικό τρόπο στα δικά μας τα κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας καθησυχάσω. Οι περισσότεροι παρόντες ε, βουλευτές καταλαβαίνουν τι σημαίνει διαρθρωτικό έλλειμμα. Προφανώς και το καταλαβαίνουν. Και τώρα να δώσω το λόγο στον συμπρόεδρό μου κύριο Γκουαλτιέρη για τη δική του παρέμβαση. Παρακαλώ κύριε Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι έχουμε σαφή συνέστηση και όπως μας κατέδειξε σαφώς και η ομιλία από το Ολλανδικό Ελεκτικό Συνέδριο το πλαίσιο διακυβέρνησής μας δεν είναι παρκές για να διασφαλίσουμε βέλτιστη διαχείριση της οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης. Άρα πρέπει να εμβαθυνθεί η ΟΝΕ και μάλιστα να αποκτήσει νέα όθηση με βάση τις καθευτήρες γραμμές τη έκθεση των πέντε πρόεδρων. Ακόμη και οι πιο φιλόδοξοι στόχοι αυτή τη έκθεση συζητιώνται αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι θετικό. Και οι πιο σημαντικοί κεντρικοί τραπεζίτέ πρόσφατα συνένεσαν προς αυτήν την ε, πορεία δημιουργία ενό Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών. Βεβαίω θα πρέπει να γνωρίζει αρκετά για αυτά τα θέματα, αλλιώ ε, θα είχαν προβλήματα. Και επίση πρέπει να έχει και τη δική τη ε, δημοσιονομική δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ίδιου πόρου. Αν θέλουμε αυτοί οι στόχοι να επιτύχουν, που είναι αναγκαίοι, αλλά που ίσω δεν είναι ακόμη εφικτοί, αν θέλουμε λοιπόν να γίνουν πιο εφικτοί, πρέπει να ξεκινήσουμε με βάση τι συνθήκε και τα μέσα που ήδη διαθέτουμε να τα αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε πολύ δυσχερείς προκλήσεις της παρούσας οικονομικής φάσης. Οπότε, διαφωνώ με τους Βάιντμαν και Μπλιγόντο Γκαγιά που λένε ότι έχουμε μόνο δύο εναλλακτικέ. Είτε θα αλλάξουμε τις συνθήκες για να υπάρξει πλήρης εχώρηση κυριαρχίας είτε πρέπει να έχουμε μια αποκεντρωμένη προσέγγιση που να βασίζεται σε ατομική ευθύνη και πιο αυστηρού κανόνες. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και τρίτη δυνατότητα και ότι έχουμε καθήκον να την αξιοποιήσουμε. Αν θέλουμε να υπάρξει απασχόληση, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στις οικονομίες μας. Και αν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα βήματα και όχι γενικές διακηρύξει προς μία ΟΝΕ. Ναι. Η Επιτροπή Γιούγκερ νομίζω ότι είναι περισσότερο υπέρ αυτού του μείγματο πολιτικών που θα βασίζεται σε πιο γενικευμένη αλλά και πιο ευέλικτη χρήση των διαφόρων δυνατοτήτων που έχουμε. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να αποκτήσει νέα όθηση και να ενισχυθεί. Γιατί είναι πολύ ακόμη ευαίσθητη η οικονομική ανάκαμψη και αντιμετωπίζουμε πολλού κινδύνου ε, στο παγκόσμιο επίπεδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που να ευνοήσει περισσότερο την ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα Πρέπει να έχουμε μια σταδιακή αλλά βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή αξιοποιώντας πλήρως την ευελιξία και πλήρως ορισμένα στοιχεία που δεν αντιμετωπίστηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν όταν αναθεωρήσαμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξη. Όπως για παράδειγμα ο χαμηλό πληθωρισμό. Επίσης κάτι πολύ σωστό που είπε η κυρία Ραμπό. Χρειάζεται απλούστευση να έχουμε περισσότερους ονομαστικούς ε, δείκτες και τιμές αναφοράς και λιγότερες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Αυτή νομίζω ότι είναι η γραμμή και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και νομίζω ότι αυτό συμβαδίζει, συμβαδίζει και με το άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Επίσης, αναφέρεται ότι τιμές αναφοράς για τις δαπάνες μπορεί να είναι ισοδύναμες με τις, ε, δημοσιο... με τις, συγγνώμη, μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως το δημοσιονομικό χώρο όσων έχουν πολλά. Το τρίτο στοιχείο αφορά την ε, σύνθεση του προπολογισμού. Πρέπει να είναι πιο ε, προσιλωμένο στις επενδύσεις. Βεβαίω χρειάζονται και διαστοτικέ μεταρρυθμίσει. Είναι αναγκαίε για να αυξηθεί η δυνατότητα ανάπτυξη. Η προσπάθεια καθορισμού τιμών αναφορά είναι ουσιοδέστατη. Και αυτό το δίκτυο των επιτροπών ανταγωνιστικότητας που ανέφερε ο κύριος Ντάιζελμπλουμ. Και αυτό είναι σημαντικό. Συμφωνώ με την προσέγγιση, λιγότερα μπορεί να καλύτερα. Και γι' αυτό προτείνουμε στα πλαίσια των, του οικονομικού κύκλου και κάποια κριτήρια σύγκληση. Είναι ουσιώδε λοιπόν να αξιοποιήσουμε πλήρω τα ισχυρά μέσα που έχουμε μέσω τη ολοκλήρωση τη ενιαίας αγορά. Να δημιουργήσουμε μια ενιαία κέφαλη αγορά και τα μέσα του σχεδίου Juncker που θα αντιμετωπίσουν ε, τις αποτυχίες της αγοράς και επίσης θα επιτύχουν πραγματική προσθετικότητα για να κινητοποιήσουμε επενδύσεις. Αν αυτή η πολιτική ακολουθηθεί αποφασιστικά και συνεπώς θα μπορέσει να βοηθήσει την εκτατική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει παράλληλα να έχουμε και ένα πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Άρα πρέπει να στείλουμε τα σωστά μηνύματα ότι θέλουμε να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και ότι θα χρησιμοποιήσουμε εφιώς τους κανόνες που ήδη έχουμε εγκρίνει και που προφανώς δεν πρέπει να αμφισβητηθούν. Οι αγορές δεν ενδιαφέρονται για θεωρητικές συζητήσεις για το σωστό μείγμα μεταξύ ε, κατανομής κινδύνων και μείωσης κινδύνων. Η αγορά θέλει να ξέρει αν ελέγχουμε την κατάσταση, αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα ή αν δένουμε τα χέρια μας επειδή δεν υπάρχει επαρκής ε, εμπιστοσύνη μεταξύ ημών. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί ο διάλογος, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη. Είναι ουσιώδες καθήκον. Και αυτό δεν είναι καθόλου μικρή σημασία καθήκον της διακυβερνητικής συνεργασίας όπως για παράδειγμα η παρούσα καθηκον τη διακυβερνητική συνεργασία, όπω για παραδειγμα η παρουσα συνδιασκεψη Σα ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι ολοκληρώνονται οι παρουσιάσεις ως εισαγωγή σε αυτή τη συζήτηση. Όλοι θίξατε πολλά ζητήματα προς συζήτηση. Μέχρι τις 11 θα έχουμε συζήτηση. Ξέρω ότι ήταν υπόμονη να πάρετε τον λόγο οι βουλευτές. Ο συνάδελφος όμως θα διαχειριστεί νομίζω αυτή τη συζήτηση, οπότε αφήνω σε εσά τη συνέχεια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι. Πρώτος ομιλητής. Από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Χόρκε Ολιβέιρα. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η έννοια έχει σημασία στις δημοσιονομικές ε, συνθήκες σε μια χώρα με προβλήματα στο έπαινε είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί η χρέωση, η δημόσια χρέωση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή και άμεση. Η εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων δεν θα έπρεπε να έχει περισσότερη σημασία στα πλαίσια της εφαρμογής των χωρών μελών γιατί όπως είπε και η κυρία Ραμπό δεν μπορούμε να μετρήσουμε καλά. Thank you. André Postema. André Postema. Κατοχώρες. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, οι διασκέψεις για το άρθρο 13 εδώ και στο Βίλνιους και στη Ρώμη και στο Λουξεμβούργο ασχολούνται με την οικονομική και δημοσιονομική κρίση και τους κανόνες της ίδιας της διάσκεψης. Ήρθε ο καιρός όμως να αλλάξουμε οπτική γωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα αισιόδεξο όργανο αλληλεγγύης που δεν δημιουργήθηκε σε εποχή χωρίς κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βασίζεται στην ειρήνη, στη συνεργασία και στην πρόοδο. Και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις διασκέψεις του άρθρου 13 για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθώ στην ποιότητα των δημοσίων δαπανών. Για τους πολιτικούς το ποσό των χρημάτων που διατίθεται για διάφορους πολιτικούς στόχους θεωρείται κάτι πιο σημαντικό από το ίδιο το αποτέλεσμα των δαπανών. Σε πολλές χώρες μέλη έχει υπάρξει πρόοδος, ώστε να μην μετράει μόνο η νομιμότητα των δαπανών, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους. Όμως, και αυτό είναι το ερώτημά μου προς το πάνελ, και κυρίως προς την κυρία Βαλερή Ραμπό, της Οικονομικής Επιτροπής ε, της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και προς τον κύριο Φεντρίκα από το Λαδικό ελεκτικό συνέδριο, Ποιε είναι οι νέε ευκαιρίε προκειμένου οι δημόσιε δαπάνε να είναι όντω επιτυχεί και αποτελεσματικές. Να έχουν αντίκτυπο δηλαδή. Και πώς θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε τέτοιες πρακτικές, όχι μόνο στην δημοσιονομική διαδικασία των χωρών μελών, αλλά και στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική διαδικασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Δημήτρης Παπαδημούλη, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι στόχοι που περιγράψατε κύριε Ντάισεμπλουμ ε, κινούνται προς μια κατεύθυνση αποδεκτή, αλλά έχω την εντύπωση ότι γίνονται πολύ αργά και πολύ λίγα σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες. Εδώ και χρόνια πολλοί κριτικάρουν την έλλειψη διαφάνειας στο πώς λειτουργεί το Eurogroup. Μόλις χθες ανακοινώσατε κάποια μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση. Είναι σωστή η ανάγκη ε, να υπάρχει εμπιστοσύνη των αγορών στις οικονομίες μας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πώς κινείται η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Και εδώ έχουμε ελλείμματα. Έχουν πέσει οι επενδύσεις, έχει μειωθεί η απασχόληση και έχει αυξηθεί η ανεργία, έχουν αυξηθεί οι ανισότητες και έχει μειωθεί η συνοχή και η κοινωνική και η εδαφική και άρα χρειάζονται περισσότερα. Συμφωνώ απολύτως ότι χρειάζονται νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, ισορροπημένα, αλλά χρειάζονται και περισσότερες επενδύσεις και περισσότερη Ευρώπη στην ενίσχυση των πολιτικών συνοχής και φορολογική εναρμόνιση έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση των φορολογικών παραδείσων και μερική αμοιβεοποίηση του χρέους. Δεν μπορεί να έχουμε μια Ευρώπη à la carte με κοινό νόμισμα και 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Με κοινό νόμισμα και 28 διαφορετικές πολιτικές για το χρέος. Η αμερικανική οικονομία έχει ανακάψει ταχύτερα από την ευρωπαϊκή γιατί εκεί δεν θεωρούν επαναστάτη τον Κέινς και την πολιτική ζήτηση. Και κάτι ακόμη. Νομίζω ότι η αναβολή για μετά το 17 των αλλαγών που χρειάζονται με ισχυρότερες μεταβιβαστικές πληρωμές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης ε, είναι λάθος. Χάνουμε πάλι χρόνο αποφεύγοντας τα προβλήματα. Ευχαριστούμε. Η Μπόκης από το Κοινοβούλιο της Λετωνίας, παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπροσωπώ το λεγκτικό συνέδριο του Λετωνικού Κοινοβουλίου. Ακούσαμε τι έχει γίνει στους Δήμους, έχουν ελεγχθεί σχετικά με τα κονδύλια. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις. Ο κόσμος όμως είναι δυσαρεστημένος. Και είναι δυσαρεστημένος γιατί υπάρχει μια μακρά διαδικασία για να βρούμε τους υπεύθυνους σε περίπτωση που υπάρχουν παραβιάσεις. Έχουμε παραβιάσεις κατάχρησης κονδυλίων. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Βέντρικ ο οποίος είναι στο ελεγκτικό συνέδριο στις κάτω χώρες. Δεν πιστεύετε ότι και σε αυτό το ζήτημα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για να βελτιώσουμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι στις χώρες μέλη η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα και χρειάζονται βελτιώσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καρέσου από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα αυτό της κατάχρησης, μάλλον συγγνώμη, το θέμα αυτό της υιοθέτηση των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Προσωπικά εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα ότι το σύστημα αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει με επιθαρχικές κυρώσεις. Αυτό απομακρύνει ακόμα περισσότερο τους πολίτες από την Ευρώπη. Συνεπώς πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, πώς δηλαδή θα αποδεχτούν σαν δικούς τους τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωζώνης. Και είναι κάτι βέβαια που προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεργαζόμαστε μαζί της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων προσπαθεί να προσαρμόσει καλύτερα τις προτάσεις της στην εθνική πραγματικότητα κάθε φορά παλιά που είχαμε συστάσει σε διάφορες χώρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε την αίσθηση ότι ήταν ίδια συνταγή για όλους, η ίδια πολιτική για όλους. Νομίζω λοιπόν ότι όντως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές ε, ιδιαιτερότητες, η πραγματικότητα στην κάθε χώρα. Και αυτό σημαίνει διάλογος και με τα εθνικά κοινοβούλια, γι' αυτό και είναι τόσο αναγκαίος. Τώρα πιο συγκεκριμένα θέλω να επιμείνω σε δύο ζητήματα. Το πρώτο το είπα και χθε. Υπάρχουν υπερβολικά πολλές διαδικασίες επίβλεψης με επικάλυψη. Επικαλύπτουν οι μεν τις δε. Και μερικές φορές αυτό οδηγεί σε συστάσεις αντιφατικέ μεταξύ τους. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει κάπως συγχώνευση του διαδικαστικού αυτού συστήματος. Διότι αλλιώς αντιλαμβανόμαστε λιγότερο καλά τις συστάσεις που γίνονται. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για το χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά τη Γαλλία, για παράδειγμα, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προπολογισμό μας έρχονται αρκετά αφού έχει αρχίσει η συζήτηση για τον προπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση. Καταλαβαίνετε είναι δύσκολο μετά να χειριστούμε τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε πρώτα να έχουμε τις συστάσεις. Μόνο τότε θα μπορούμε να τις καταλάβουμε και καλύτερα και να τις αποδεχτούμε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Σημαντικό αυτό που είπατε. Άλπερτ Σαν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν βλέπω το Μπερές. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την συνεδρίαση αυτή που πραγματικά βρίσκεται στο κέντρο αυτού που θα έπρεπε να είναι η διάσκεψη 13. Μπαίνουμε δηλαδή στην καρδιά της συζήτηση σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια και βλέπουμε ότι αυτή η διτή προσέγγιση είναι αναγκαία αν θέλουμε να δώσουμε ε, σημασία στον συντονισμό των οικονομικών μας πολιτικών. Τρεις παρατηρήσεις έχω. Πρώτον, ο πρόεδρος Τάισελμπλουμ έχει προδεύσει στο θέμα της διακυβέρνησης του Eurogroup, τον ευχαριστώ και τον συγχαίρω γι' αυτό. Βέβαια θα πρέπει να πάμε ακόμα περισσότερο, πιο πέρα. Αν ε, θέλουμε να υπάρχει μια ολοκλήρωση στην ε, Ευρωζώνη, άρα η διάστρωση ανάμεσα στην κοινοτική μέθοδο και τη λειτουργία του Eurogroup μας ε, οδηγεί σε μαθήματα, ιδίως ε, αν λάβουμε υπόψη μας τις μακρές διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. Άρα ίσως υπάρχουν ακόμα προοπτικές εξέλιξεις και βελτίωσεις στο μέλλον και σύντομα θα έλεγα. Τώρα θέλω επίσης να ευχαριστήσω πολύ τον Κες Φεντρίκ για αυτό που είπε. Για δύο πράγματα κυρίως. Πρώτα απ' όλα γιατί είπε ότι δεν πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια οικονομική διακυβέρνηση που να βασίζεται μόνο σε κανόνες. Όντως δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε κανόνες γιατί αυτό μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Κάτι το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε και ακριβώς αυτό προσπαθούμε. Τον ευχαριστώ επίση που είπε ότι έχουμε ένα σωρό εργαλεία τα οποία όμως δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως. Η διαδικασία λοιπόν διαπίστωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών, για να το πω έτσι κάπως κομψά, μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Και έτσι έρχομαι σε δύο προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση την οποία ετοιμάζουμε ως συστάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Και στην έκθεση αυτή υπάρχουν δύο άξονες που θέλω να αναφέρω. Ο ένας είναι η χρήση των συστάσεων για την Ευρωζώνη, που πρέπει να καταλήξουν στην αρχή του κύκλου να έχουμε στόχους για την Ευρωζώνη σε επενδύσεις. Ακριβώς γιατί κάποιοι κανόνες έχουν προκυκλικό χαρακτήρα και άρα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις. Και δεύτερον, πάλι στην αρχή της διαδικασίας, να υπάρχει ένας κώδικα συντονισμού που να επιτρέπει ένα πολιετές πρόγραμμα γύρω από στόχους που να βασίζονται στο θεματολόγιο 2020. Δεν έχω χρόνο να αναπτύξω, αλλά καλύτερη χρήση των συστάσεων και κώδικας συντονισμού. Ευχαριστώ. Τώρα πρέπει να επιμείνουμε στα δύο λεπτά, έτσι. Πρέπει πειθαρχία για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους όσους το ζήτησαν. Επόμενος ομιλητής, Sir William Cash, από την Βουλή Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι επειδή δεν είμαστε στην Ευρωζώνη, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε αυτό το πλαίσιο, αλλά βεβαίως και εμάς μας επηρεάζουν τα όσα συμβαίνουν. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω και υπάρχει και το θέμα του δημοψηφίσματος για το κατά πόσον θα παραμείνουμε ή θα αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στα έγγραφα τα οποία μας δώσατε, διότι νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία του θέματος. Παραδείγματο χάρη, ναι, το γεγονός ότι δεν υπήρχαν επαρκείς μηχανισμοί προσαρμογής για να αντιμετωπίσουν τα σύμμετρα σοκ. Ε, σίγουρα όλο αυτό αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά αναφέρεται ε, ο συντονισμό των εθνικών οικονομικών πολιτικών που αποδείχθηκαν ε, ανεπαρκεί. Και μετά στη συνέχεια λέει ότι τα θεσμικά όργανα επάσχουν από δημοκρατικό έλλειμμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Και με δύο λόγια, και μόνο αυτό θέλω να πω, είναι αυτά που άκουσα από τι ε, εκθέσει και τι παρουσιάσει πρόκειται για μία αύξηση προ ένα ε, σύστημα ελέγχων και διαταγών, το οποίο πόρο απέχει από το δημοκρατικό έλεγχο και εμείς στο Westminster από το 17ο αιώνα και μετά εργαζόμαστε στη βάση μιας κυριαρχίας η οποία σχετίζεται επακριβώς με το θέμα της φορολόγησης και των δαπανών. Το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη το 2004 το έφερε η Γερμανία κλπ. Το θέμα είναι κατά πόσον ε, ε, η Ιταλία αυτή τη στιγμή τη διατάζουν τι να κάνει. Και πρέπει λίγο να δούμε και τη σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών. Το αρχιτεκτονικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Τα εθνικά κοινοβούλια κατά την άποψή μα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του ζητήματο, όπω είπε και ο Ντέιβιτ Κάμερον στην ομιλία του στον Γκρούμπερτ. Και επίση πρέπει να σα πω ότι δεν θεωρούμε και εμείς και οι φίλοι μου ότι πηγαίνει αρκετά μακριά στις διαπραγματεύσεις και πρέπει να αποχωρήσουμε γιατί αυτά τα θύματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Διακόπτει ο Πρόεδρος, ο κύριος Γεράσιμος Μπαλαούρας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ε, Ελλάδα έχουμε μια παροιμία που λέει «Ή ο στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Και εδώ το δεύτερο ισχύει για, νομίζω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωζώνη. Υπάρχει το σύμφωνο της σταθερότητας, το οποίο είναι ένας κορσές στην ανάπτυξη. Και μάλιστα ένας κορσές που άλλοι το φορούν πολύ στενά και άλλοι πολύ χαλαρά, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, που είχαν μια άλλη μεταχείριση. Σήμερα άκουσα από εισηγητές πανηγυρικούς τόνους ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι, έχουν μια σήμαντη αύξηση του 0,9%. Μα μπορούμε άραγε να βγούμε από τη βαθιά ύφεση με τέτοιες θέσεις. Είναι αντιγραφή των θέσεων του Δούνου του, η οποία, το οποίο έχει καταγράψει ιστορική αποτυχία όπου εφάρμοσε αυτές τις συνταγές. Και έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα και όχι μόνο στη χώρα μου, στην Ελλάδα, που εκεί είναι τραγικά τα πράγματα εξαιτία των πολιτικών αυτών, έχουμε ύφεση βαθιά, έχουμε ανεργία, έχουμε φτώχεια, έχουμε να χάσιμο των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Και μάλιστα επιπλέον ότι στην Ελλάδα τριπλασιάστηκε το χρέος από την, ε, την πεταετία που πέρασε λόγω της εφαρμογής της σκληρής πολιτικής λιτότητας και για να εξηγηθούμε. Άλλο συνετή διαχείριση και άλλο κορσές της ύφεση. Η για παράδειγμα αγαπητοί συνάδελφοι οι Ηνωμένε Πολιτείε μπήκαν σε ύφεση την ίδια εποχή που μπήκαμε και εμείς. Είναι τώρα δυόμιση με τρία χρόνια που έχουν ανάπτυξη. Δεν μας προβληματίζει άρα γι' αυτό. Ακόμα όμως και η επιστοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Συνάντηση κόντρα από πολλέ. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Κάναμε... Τελειώνω. Ε, θέλουμε και επενδύσει, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, που οι οποίε θα έχουν στρατηγική και θα είναι ψίχουλα. Ευχαριστώ κύριε. Mr. Ο κύριος Σόμπορ από την ε, Ουγγρική Εθνική Συνάδελφος. Η κυρία Σόμπορ. Από το 2011 τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν αναπτύξει διάφορες πρακτικές για την οικονομική διακυβέρνηση. Στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στα θέματα αυτά. Προσαρμόζουμε το θεματολόγιό μας ε, στα πιο σημαντικά γεγονότα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και συζητούμε βασικά στοιχεία οικονομικής ε, πολιτικής και συντονισμού και ε, οι αρκετές φορές έχουμε παρουσιάσει την άποψή μας. Η πιο πρόσφατη συνεδρίασή μας έγινε το Δεκέμβριο πέρσι. Συζητήσαμε τα έγγραφα τα οποία δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Νοεμβρίου και αναθεωρήσαμε και την εμπειρία των προηγούμενων πέντε ευρωπαϊκών εξαμήνων. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω λοιπόν τη θέση της Ουγγαρίας ε, σε όλα αυτά. Συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με τις βασικές προτεραιότητες ε, της έκθεσης ανάπτυξης και της επενδύσεις ε, στην Ουγγαρία για το μηχανισμό τάκτου ανάγκη. Ωστόσο θεωρούμε ότι κάτι λείπει και λείπουν δηλώσει για την εφαρμογή του αρχικού στόχου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την εφαρμογή του Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ε, καλωσορίζουμε τον εξορθολογισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την απλούστευμένη και μικρότερη εκδοχή των συστάσεων αναχώρα. Όσον αφορά τις συστάσεις αυτές, ε, πιστεύουμε ότι χρειάζεται να αφιερώνεται περισσότερο χρόνος στη συζήτηση επί ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και ε, την εφαρμογή στα κράτη-μέλη αυτών των συστάσεων. Οι συστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν γενικούς ε, πολιτικούς στόχους και δεν θα πρέπει να περιγράφουν και να συνταγογραφούν συγκεκριμένα μέτρα. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται αρκετό περιθώριο ευελιξίας για να μπορέσουν να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία πολιτικής πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα συνεισφέρουν στην ε, ε, επιτυχή εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα. Ολοκληρώνοντας, ε, θα ήθελα να σας πω ότι οι φετινές συστάσεις αναχώρα ελπίζουμε να αντακατοπτρίζουν μια σωστή εικόνα για τις οικονομικές προοπτικές της Ουγγαρίας. Ο κύριος Γιωακίμ Μπός από το Γερμανικό Κοινό. Yeah. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκε κάτι που έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα. Σε πολλές χώρες η ανταγωνιστικότητά μας αντιμετωπίζεται από τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Πρέπει να καταλάβουμε πώς είναι, σωστές, πώς είναι η σωστή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στις χώρες αυτές, γιατί για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την έλλειψη εμπιστοσύνη από του έντιμου φορολογούμενου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει σήμερα να αναφερθεί. Και σε σχέση με αυτό, να κάνω μια ερώτηση συγκεκριμένα στον κύριο Ντάιζελμπλουμ. Προτίθεται η Ολλανδική Προεδρία και κυβέρνηση να σκεφτεί πώς μπορεί με το δικό της υπόδειγμα, με την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής η οποία γίνεται εις βάρος των εντύμων φορολογούμενων και των εντύμων επιχειρήσεων. Προτίθεται λοιπόν η Ολλανδική κυβέρνηση να κάνει κάτι για να μην υπάρχουν αυτές οι ειδικέ ρυθμίσεις που στην ουσία είναι φορολογικό dumping της Ολλανδίας σε βάρος των άλλων. Προτίθεται να κάνει κάτι συγκεκριμένο για να το καταπολεμήσει αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Φρατσέσκο Καριέλο, Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας παρουσιάσω την ιταλική εμπειρία εδώ. Η Ιταλία εισήγαγε τον ισοσκελισμένο προπολογισμό μετά από το θέμα του Δημοσιονομικού Συμφώνου το 2012, αλλά στην πράξη ανέστηλε τρεις φορές την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου, ο οποίος ε, αυτή τη στιγμή είναι για το 2018. Να σας πω δηλαδή ότι με βάση αντικειμενικά στοιχεία το δημοσιονομικό σύμφωνο δεν οδηγεί σε καμία ανάπτυξη στη χώρα μας, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό αποδεικνύεται αντίστοιχα με τα ίδια αντικειμενικά στοιχεία και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ το χρόνο μου για να σας πω ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του ε, Δημοσιονομικού Συμφώνου και του σχετικού συμβουλίου εντείνει το δημοκρατικό έλλειμμα που δημιούργησε η Ευρώπη και εσείς στον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών. Εμείς θεωρούμε ότι μια ακόμα ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη λιτότητα που συστήνεται με αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αυξήσει απλώς ε, την ε, ε, καθυστέρηση στην ανάπτυξη που υπάρχει στη χώρα μου και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς ε, να ε, ληφθεί η γνώμη των, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία ελήφθη αυθαίρετα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα εδώ, κατά την άποψή μου, να ε, δώσουμε περισσότερες εξουσίες τη δική μας την κοινοβουλευτική συνέλευση να εκφράζουν την άποψή τους στο Εθνικά Κοινοβούλια τουλάχιστον ως προς τον τρόπο επιλογής ε, των Συμβουλίων για τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών. Είμαστε, πρέπει να ολοκληρώσετε λέει ο Πρόεδρος, είμαστε αντίθετοι αλλά θεωρούμε ότι αν ε, υπάρχει ένα τέτοιο συμβόλαιο πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Έρικ Φαρουμέη από το Βελγικό Κοινοβούλιο. Πρόεδρε. Εδώ πρέπει να αντιμιλήσω κατά κάποιο τρόπο, γιατί στις συζητήσεις που κάνουμε εμείς για τον προϋπολογισμό έχουν γίνει πολύ περισσότερες για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή από ό,τι τελικά ο προϋπολογισμός για διάφορους τομείς. Στο Εθνικό Κοινοβούλιο συζητούμε πολύ για τον προπολογισμό. Το Βέλγιο, βλέπετε, είναι μια χώρα που ήταν κάτω από το 3% αλλά με τη χρέωση και τα λοιπά έχουμε φτάσει σε 7%. Στα εθνικά κοινοβούλια καταλαβαίνουμε ότι έχουν γίνει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με διάφορες χώρες και το Βέλγιο καταλαβαίνει ότι πρέπει να φτάσει σε ισορροπία το 2018 στον ονομαστικό προπολογισμό δε το 2019. Είναι δύσκολο και σημαίνει 1% το χρόνο πρέπει να μειώσουμε το χρέος. Όλοι λένε ότι είναι δύσκολο αυτό να επιτεθεί. Οι συμφωνίες λοιπόν που επιτυχάνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του συμφώνων Ανάπτυξης και Σταθερότητας πρέπει να αναθεωρηθούν. Διότι λέμε περισσότερα χρήματα να δώσουμε για την ασφάλεια, για το άσυλο, για το προσφυγικό. Η οικονομική ανάπτυξη τελικά μένει πίσω και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει βοηθήσει όσο θα έπρεπε την πραγματική οικονομία και οι επενδύσεις σίγουρα είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι θα έπρεπε. Πολλά επιχειρήματα λοιπόν υπάρχουν για να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της την πραγματική οικονομική κατάσταση και τις δαπάνες που γίνονται για τους πρόσφυγες από την κάθε χώρα κλπ. Και να ξαναδούμε το θέμα των κανόνων για τα ελλείμματα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Καλή ερώτηση. Ευχαριστούμε. Ρίτα Μίλλερ. Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στη Φιλανδία, το κοινοβούλιο μας Καταρχήν, κατευθύνει πάρα πολύ καλά το κοινοβούλιο μας, όταν, ε, την κυβέρνησή μας, όταν η κυβέρνηση ε, λαμβάνει θέση και τοποθετείται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κατά την άποψή μας όμως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, συγγνώμη, είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε πολύ καλά στο Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Και οι πολίτες δεν γνωρίζουν το ζήτημα. Δεν ε, ε, είναι εξοικειωμένοι με το ζήτημα. Επομένως, καλό είναι να έχουμε και τις συμβουλές σας και την άποψή σας για το πώς μπορούμε ε, να αναπτύξουμε και αυτή την πλευρά. Για μας είναι ζωτική σημασία όταν συζητούμε για τα κοινά οικονομικά μας και λαμβάνουμε αποφάσεις εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αποφάσεις αυτές ε, να επιχειρώνονται και από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν ακούσει τους ε, εθνικούς οργανισμούς, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, ώστε να διαβιβάζονται και οι απόψεις των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε προχωρήσει σε απλούστευση και στις διαδικασίες και ε, έχουμε βελτιώσει και το χρονοδιάγραμμα, διότι αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συνεισφέρουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επίσης θεωρούμε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι λέγεται ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να είναι στη διάρκεια μιας κυβερνητικής θητείας, όχι μια ετήσια διαδικασία. Ε, ελπίζω λοιπόν, και εδώ έρχεται και η ερώτησή μου, Όταν σκεφτόμαστε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα ώστε να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από τις εθνικές αποφάσεις. Ο κύριος Κουράκης, Ελληνικό Κοινό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ασχοληθεί με το πρόβλημα της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέοι θεσμοί έχουν συσταθεί, πολύπλοκοι μηχανισμοί της οικονομικής διακυβέρνησης έχουν τεθεί σε λειτουργία και ένα μεγάλο μέρος της εθνικής κυριαρχίας σε σχέση με την οικονομία έχει μεταφερθεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Συνεχίζονται διαπραγματεύσει σχετικά με του προπολογισμού και του μηχανισμού οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχουν λάβει χώρα, αλλά θα μπορούσε κανεί να πει βάσιμα ότι όλο αυτό το σύστημα δεν χαρακτηρίζεται ούτε από διαφάνεια, ούτε σε ορισμένες περιπτώσεις από αποτελεσματικότητα. Τα γεγονότα αυτά οδηγούν σε μια ενοποιημένη εικόνα μιας οικονομίας σε βαθιά κρίση, ευάλωτη στην κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών και αυτό τελικά οδηγεί σε απώλεια της πολιτικής νομιμοποίησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Το οικονομικό περιβάλλον στις ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνεται εχθρικό λόγω των συνεχών φόρων και η κοινωνική προστασία έχει καταρρεύσει ενώ οι κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης που επιβάλλονται κινούνται στη λογική της εξουσίας. Αυτό το μοντέλο έχει αποτύχει, μεν, αλλά εξακολουθεί να μην αλλάζει. Όταν ορισμένες κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προτιμούν τελικά το μονοπάτι που επιβάλλουν οι αγορές. Και στο τέλος, η αποτυχία των αγορών οδηγεί σε μια νέα αποτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο δημοκρατικός έλεγχος είναι πολύ περιορισμένος σε όλες αυτές τις διαδικασίες ο έλεγχο των εκλεγμένων οργάνων στη διαδικασία λήψη αποφάσεων στην οικονομία είναι εξαιρετικά αδύναμο. Οι γνώμε των Εθνικών Κοινοβουλίων δεν λαμβάνονται υπόψη σοβαρά. Τα μόνο κριτήρια που επιβάλλονται είναι από τι αγορέ. Θα ήθελα να πω ότι η γνώμη των πολιτών δεν λαμβάνεται υπόψη και αυτό έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών, όταν κάθε δημοψήφισμα για το μέλλον τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είχε αρνητική έκβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γαλλία, στην Ορβηγία, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, για στον ανθρώπο. Next speaker, Baroness. Ευχαριστώ. Η Βαρόνη Φόρτνερ από την Βουλή των Λόρτων στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να καθησυχάσω τις συναδέλφους ότι δεν υπάρχει μόνο μία άποψη για την παραμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ νομίζω προσωπώ την άλλη άποψη. Θέλω λοιπόν να γίνει διαπραγμάτευση και να δώσουμε μια μάχη για να κερδίσουμε. Θα ήθελα να συνεχίσω από αυτά που είπε ο κύριος Βλούμ για το τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν στις ε, συστάσεις αναχώρα. Πιστεύω ότι είναι εύρωστε οι προτάσει του ότι θα πρέπει να γίνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά θα ήθελα να σταθώ στο θέμα τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Εχθέ έγινε μια συζήτηση για την επέκταση των δικτών στο πίνακα βαθμολόγηση ε, και μου φαίνεται ότι αυτό στην πραγματικότητα έρχεται να χτυπήσει άντρα σε αυτό που θέλετε από αυτές τις συστάσεις ανά χώρα. Ή θα το αφήσετε στη χώρα και στους μηχανισμούς εποπτείας της, όπως για παράδειγμα στο Κοινοβούλιο, ή θα το επιβάλλετε κεντρικά. Και τα επιχειρήματα, ε, από ό,τι φαίνεται σήμερα, πηγαίνουν κατά της κεντρικής ε, επιβολής. Εμείς ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαβουλευόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους αυτούς καθεαυτού. γίνεται όμω μια διαβούλευση, γίνεται μια εκτίμηση επιπτώσεων, ε, υπάρχουν διάφορε ομάδε πίεση και υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι και αρκετέ ισορροπίε για να μπορέσει ο καθένα να τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση. Και θεωρώ ότι το να θέλουμε να έχουμε κεντρικά τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των κοινωνικών δεκτών είναι προ τη λανθασμένη κατεύθυνση. Και επειδή δεν έχω και αρκετό χρόνο, θα ήθελα να ρωτήσω την εξή ερώτηση και όποιο θέλει να την απαντήσει. Την έθεσε και χθε. Η Ευρωζώνη πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να υπάρχει ένας Υπουργό Οικονομικών της Ένωσης. Υπήρχε στην έκθεση των πέντε προέδρων, αγνοήθηκε ε, και ε, όλο ανακύπτει το ζήτημα αυτό. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να μας πείτε κατά πόσον θεωρείτε ότι χρειάζεστε έναν Υπουργό Οικονομικών. Ο κύριος Παόλο Περέιρα τώρα από την ε, Πορτογαλική Βουλή. Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι η Πορτογαλία κάνει τη δουλειά της και σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής. Σε θεσμικό επίπεδο έχουμε ε, συστήσει ένα δημοσιονομικό συμβούλιο το οποίο αναλύει τον προπολογισμό και τις μακροοικονομικές προβλέψεις και έχουμε και ένα τεχνικό τμήμα για την υποστήριξη του προπολογισμού στο Κοινοβούλιο που ε, εργάζεται για την αρμόδια επιτροπή και αναλύει και ανεξάρτητα για κάθε πολιτικό κόμμα τον προπολογισμό. Έχουμε λοιπόν τους κατάλληλους θεσμούς, ε, προσπαθούμε να μειώσουμε το έλλειμμα του ΑΕΠ, να σταθεροποιήσουμε το ΑΕΠ ε, ακόμα βέβαια έχουμε κάποια προβλήματα. Επομένως αυτό το πρώτο τμήμα της παρέμβασής μου θα πρέπει να πω είναι για να πω ότι τηρούμε τους κανόνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την ε, διακυβέρνηση ε, του οικονομικού και δημοσιονομικού συμφώνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτησή μου απευθύνεται προ τον κύριο Μπλουμ και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον ξέρετε οποιαδήποτε ένωση νομισματική στην Ένωση που να μην έχει και μία ένωση ε, δημοσιονομική που μπορεί να απορροφήσει τα σύμμετρα σοκ στα κράτη-μέλη. Και επειδή η απάντηση φαντάζομαι ότι θα είναι αρνητική, τι συγκεκριμένα βήματα θεωρεί το Eurogroup ότι πρέπει να ληφθούν για να έχουμε αυτή την ένωση. Διότι έχουμε ένα προϋπολογισμό 1%, 1 του ΕΟΠ, το 84% δεν είναι στη διακριτική μας ευχαίρεια, επομένως δεν έχουμε καν τη δυνατότητα να ταπανίσουμε κάποια επιπλέον κονδύλια για τους πρόσφυγες, γιατί τα πάντα είναι καθορισμένα συγκεκριμένα που θα πάνε. Με αυτό λοιπόν το μοντέλο πολύ δύσκολο μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ μακριά με το ευρώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλφρετ Σάντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι τονίζουμε την ανάγκη να υπάρχουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο για να μπορέσουμε να έχουμε ανάκαμψη. Μας λένε συνεχώς ότι με την ολοκλήρωση των δημοσίων ε, προπολογισμών και με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις θα ακολουθήσουν οι επενδύσεις. Όπως έγραψε ο Ρέντσι στη Λα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Οι πολιτικοί λιτότητες δεν έχουν οδηγήσει σε ανάπτυξη και θέσει εργασίας, κάθε άλλο. Και μάλιστα στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου δεν είχαμε ε, λιτότητα στο επίκεντρο, έχουμε ανάπτυξη και θέσει εργασίας. Όποια ανάπτυξη έχει υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται στη μείωση των τιμών του πετρελαίου, στην ποσοτική χαλάρωση και στην στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα και όχι μεγαλύτερες επενδύσεις. Επίσης μπορεί να έχει συνεισφέρει και σε πληθωριστικές τάσεις οι οποίες δεν θα επιτρέψουν νέες επενδύσεις. Θα συνεχίσουμε να καθυστερούμε λοιπόν σε νέες επενδύσεις και σε δημόσιο αλλά και μετά θα ακολουθήσουν και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις καθυστερούν και εάν οι δημόσιες επενδύσεις δείξουν ότι υπάρχει ανάπτυξη ε, μόνο έτσι έχουμε ιδιωτικέ επενδύσει. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερε δημόσιε επενδύσει σε οικονομικέ υποδομέ, ε, στην παιδεία, στην προώθηση τη εκβιομηχάνηση, παρά το γεγονό ότι αυτό το λέμε συνεχώ, σε τομείε όπω η στέγαση, στέγαση ε, και σε άλλου τομεί. Αλλά ε, προχωρούν πάρα πολύ αργά οι δημόσιες επενδύσεις. Το είπα και πέρσι κατά τη συνεδρίαση αυτή με τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα το επαναλάβω. Οι κανόνες λειτουργίας του Δημοσίου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ δαπανών και επενδύσεων στον προπολογισμό και όλα έχουν την ίδια βαρύτητα όταν υπολογίζουμε ελλείμματα και δαπάνε. Ω αποτέλεσμα, οι κανόνε που υποτίθεται ότι μπορούν να βοηθήσουν στην εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών, στην πραγματικότητα πιέζουν τι κυβερνήσει να κόβουν τι επενδύσει για να ε, συνεχίσουν τι δαπάνε. Διακόπτει ο Πρόεδρο. Δύο τελευταίοι ομιλητέ τώρα. Ένα λεπτό ο καθένα, παρακαλώ. Μαρκ Φρανσουά από τη Γαλλική Γερουσία πρώτα. Ευχαριστώ και καλημέρα. Έχω μία ερώτηση όσον αφορά τους προσανατολισμούς έτσι όπως προβλέπονται στην έκθεση των πέντε προέδρων σχετικά με την παραγωγικότητα. Γιατί η έκθεση αυτή των πέντε προέδρων αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η δημιουργία για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών μειώνει κάποια προβλήματα, τα λύνει, αλλά ότι μένουν πολλά ακόμα να γίνουν και προβλέπει σε κάθε χώρα τη δημιουργία μιας αρχής ανταγωνιστικότητας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δημιουργία ενός οργανισμού όπου θα συμμετείχαν όλες αυτές οι εθνικές αρχές ανταγωνιστικότητας. Παραγωγικότητα λοιπόν. Οπότε οι ερωτήσεις μου είναι εξής. Πρώτον, χρειάζεται ή όχι να υπάρξει άλλο ένα τέτοιο τεχνικό όργανο, ενώ σίγουρα σε όλες τις χώρες υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις. Και δεύτερον, δεδομένων των εμπειριών που αναφέρει η εκτίση των Προέδρων Βέλγιο και κάτω χώρες όπου υπάρχουν τέτοιες αρχές, μπορούν να έχουν περισσότερες διευκρινήσεις για το πώς λειτουργούν αυτές εκεί. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μανουέλ Ροντρίγκες. Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σχολιάσω κάποια από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν για τον προπολογισμό. Επικεντρωνόμαστε στους περιορισμούς, το ρυθμό μείωσης των διευθυντικών ελλημάτων. Για πολλές χώρες μέλη δεν είναι το κύριο πρόβλημα αυτό. Το κύριο πρόβλημα είναι η μείωση του δημόσιου χρέους. Πέρα από το 5% το χρόνο. Αυτός ο υπολογισμό όμως είναι απλός και επιταχύνει απλώς την μείωση του δημοσίου χρέους, κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασία βέβαια για να μειωθεί το χρέος μιας χώρας και είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να υπάρξουν και πάλι επενδύσεις. Γιατί επικεντρωνόμαστε μόνο σε έναν κανόνα που έχει να κάνει με το σεβασμό του δημοσιονομικού συμφώνου, που είναι ο πιο απαιτητικό κανόνα, ενώ υπάρχει και ένα άλλο πιο απλό, ο οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Τώρα, να απαντήσει το πάνελ στα διάφορα σχόλια. Πρώτο, Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο. Πολλά, πολλές ερωτήσεις υπήρξαν για μένα. Πόσο χρόνο μου δίνετε, τρία λεπτά. Ωραία, η συζήτηση κλειδί εδώ έχει να κάνει με το μέλλον της διακυβέρνησης, έχει να κάνει με τον τρόπο που σχεδιάζεται. Έχουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένους κανόνες που πηγαίνουν από το κέντρο προς τις χώρες και από εκεί και πέρα είναι ευθύνη κατά πρώτον των χωρών μελών να συμμορφωθούν με τους κανόνες αυτούς. Οι κανόνες μπορεί να είναι σωστοί, μπορεί να είναι περίπλοκοι, πρέπει να τους κάνουμε πιο αποτελεσματικούς, περισσότερο κατανοητούς για τους πολίτες μας, ναι. Αλλά έτσι λειτουργούμε τώρα. Οπότε η πραγματική ευθύνη για τις αποφάσεις όσον αφορά τους προπολογισμούς, τις μεταρρυθμίσεις, πώς σχεδιάζουμε το συλλογικό σύστημα, είναι εθνική αρμοδιότητα. Και αυτό το λέω γιατί κάποιοι σήμερα είπαν ότι τα προβλήματά μας οφείλονται στο σύμφωνο σταθερότητας. Όμως, τα κύρια προβλήματα στις χώρες μας οφείλονται σε κακές εθνικές πολιτικές, λέω εγώ. Δεν έχουμε χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά διμερώς ευχαρίστως να το συζητήσουμε όσο θέλετε. Κατόπιν τούτων, μπορείτε βέβαια να το πάρετε και ανάποδα, να πείτε δεν λειτουργεί το σύστημα γιατί έχουμε αυστηρούς κανόνες, αλλά να, ο κύριος Βεντρίκ είπε ότι αγνοούνται οι κανόνες αυτοί, δεν εφαρμόζονται δηλαδή. Εντάξει, εγώ θα έλεγα σε ένα βαθμό, αλλά πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, μειώνουμε ελλείμματα, μειώνουμε το χρέος, αρχίζουμε να δημιουργούμε επενδύσεις κλπ. Οπότε εγώ είμαι κάπως περισσότερο αισιόδοξο. Αλλά όντως έχουμε αυτό το μοντέλο που βασίζεται σε κανόνες και μετά αποφασίζουν τα κοινοβούλια. Δεν λειτουργεί λέμε. Ωραία, τότε τι να κάνουμε. Κεντρική διακυβέρνηση να αναλάβουμε εγώ, εμείς τις ευθύνε στο κέντρο. Όταν όμως μιλάμε για δημοκρατική νομιμότητα και στήριξη από το κοινό, ε, δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο. Και γιατί το λέω, γιατί αν αυτές τις αρμοδιότητες τις αναθέσετε στο κέντρο, για παράδειγμα το σχεδιασμό των μελλοντικών συνταξιδοτικών μα συστημάτων, φανταστείτε να αποφασίζονται εδώ στις Βρυξέλλες ή τα συστήματα περίθαλψης, το κοινωνικό μοντέλο στις διάφορες χώρες όπου σήμερα είναι διαφορετική η κατάσταση στις χώρες ΜΕΛ. Φανταστείτε να τα αποφασίζουν όλα αυτά οι Βρυξέλλες, αναπόφευκτα γιατί αυτές είναι οι αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν τελικά πώς θα λειτουργήσουν στο μέλλον οι οικονομίες μας και πώς ο προπολογισμό μας θα είναι, θα είναι βιώσιμος. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι όταν λέμε θέλουμε περισσότερη διακυβέρνηση στο κέντρο, είναι ένα σύστημα κανονισμών που αναθέτει αρμοδιότητες στις χώρες μέλη, αν δεν λειτουργούν, αν δεν λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα, πού πάμε. Εγώ ε, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει εξέλιξη στην νομισματική ένωση. Μπορείτε να διαφωνήσετε, αλλά εγώ έτσι πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει να προχωρήσουμε για να μην χάσουμε τη στήριξη του κενού και να μην παίρνουμε ε, μεγάλες και πολλές αρμοδιότητες από τα εθνικά κοινοβούλια και να τις μεταφέρουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Τώρα για τα συμβούλια αυτά ανταγωνιστικότητα. Εντάξει, λέτε ότι έχουμε ήδη κάποιε τέτοιε αρχέ. Εντάξει, σωστά. Αν όμω την ευθύνη την αφήσουμε στο εθνικό επίπεδο, τότε α μιλήσουμε για τι εμπειρίε μα, α τι μοιραστούμε μεταξύ μα. Εγώ θέλω καλύτερο σχεδιασμό και καλύτερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ναι, απαιτεί και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Πώς θα οργανωθεί αυτό, εγώ νομίζω ότι θα οργανωθεί σε εθνικό επίπεδο. Ο κοινωνικός διάλογος δηλαδή πρέπει να γίνεται κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά στις κατοχώρες έχουμε εμπειρίες γιατί έχουμε τέτοια συμβούλια παραγωγικότητας και έχουμε συνομιλίες με τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Έχουμε εμπειρίες και με τα Συμβούλια ανταγωνιστικότητα λοιπόν είναι το κεντρικό γραφείο σχεδιασμού όπως το ονομάζουμε στις κάτω χώρες. Αυτοί όμως μας λένε σε εμά τους πολιτικούς, τέλος πάντων μας συμβουλεύουν πώς να σχεδιάσουμε τις μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους. Αν έρθουμε με κακά σχέδια, μας το λένε ότι είναι κακά σχέδια ότι θα πλήξουν την ανταγωνιστικότητά σας, την απασχόληση κτλ. Το αντίστροφο θα ήταν καλό. Χρειαζόμαστε λοιπόν βοήθεια για το σχεδιασμό των πολιτικών μας. Και δεν σας λέω ακολουθήστε το παράδειγμα των κάτω χωρών, λέω απλώ ότι πρέπει να σχεδιάζουμε καλύτερα τις μεταρρυθμίσεις μας. Γιατί αν θέλουμε να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα. Χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες πολιτικές που να μας προστατεύουν την ευημερία μας, η οποία όντω είναι μια ήπειρος ευημερούσα η Ευρώπη σήμερα με ένα καλό κοινωνικό μοντέλο. Πρέπει να τα διατηρήσουμε και τα δύο. Και τη διαφάνεια και ένα ισχυρό κοινωνικό μοντέλο. Θα απαντήσω τώρα σε μία ερώτηση από τον κύριο Γιωχήμ Πώς, ο οποίος αναφέρθηκε στη φοροδιαφυγή. Εγώ προεδρεύω τώρα στο ΕΚΟΦΗΝ έχουμε στην ημερήσια διάταξη τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, τι κάνουν οι κάτω χώρες, εγώ δεν έρχομαι εδώ σαν Ολλανδός υπουργό, αλλά αφού με ρωτήσατε, απαντάω έτσι. Συμφωνήσαμε με τη Γερμανία να ανταλλάξουμε τα... τους κανόνες μας όσον αφορά το θέμα αυτό της φοροδιαφυγής. Εντάξει, ό,τι θέλετε, όλες τις διευθετήσεις φορολογικές που κάνουμε εμείς, θα σας τις δώσουμε και είμαστε πολύ, θέλουμε και εμείς πολύ να ξέρουμε τι κάνουν οι Γερμανοί με τις δικές τους επιχειρήσεις. Έπειτα, να δούμε τις διάφορες συμφωνίες που υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει να αποφεύγουμε τη διπλή φορολόγηση. Αλλά να μην υπάρχει βέβαια και διπλή έλλειψη φορολόγησης, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οπότε θα αλλάξουμε τις συμφωνίες. Έπειτα, εμείς ως Ολλανδική Προεδρία πιέζουμε σε αυτό το εξάμεινο να υπάρξει πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρειάζομαι και τη δικιά σας στήριξη, της Γερμανίας δηλαδή. Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να δεχτούν το συνολικό πακέτο και μην αρχίζουν τα παζάρια. Ε, μην λέμε θέλουμε περισσότερο χρόνο. Εντάξει, όλοι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Ελπίζω λοιπόν να το πετύχουμε αυτό το εξάμεινο με τη στήριξη και της δικιάς σας κυβέρνησης, της Γερμανικής. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Κις Φέντρικ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, στην επαγγελματική μου, με την επαγγελματική, του, επαγγελματική μου ιδιότητα είμαι πολύ μετριόφρον. Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να απαντήσω στην ερώτηση πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για δημοσιονομικά θέματα. Ναι, είναι σωστό ερώτημα. Και υπάρχουν πολλές απαντήσεις να αναφέρω δύο ενδεχομένε. Να διορθώσουμε τα λανθασμένα συστήματα για δαπάνες. Για παράδειγμα, πολλά δις που συλλέγει η κεντρική κυβέρνηση μέσω φορολογία δίδονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για συγκεκριμένες ε, υποδομές και τα λοιπά και δαπάνες. Αλλά από πλευράς αποτελεσματικότητας είναι κακό αυτό το σύστημα γιατί το μόνο που ενδιαφέρει τους ε, ΟΤΑ είναι να τα δαπανίσουν όλα. Και το ερώτημα τι η αξία παράγεται για τους πολίτες μέσω των χρημάτων των φορολογουμένων είναι κάτι που είναι δευτερεύον για αυτού. Αν θέλετε λοιπόν να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση για το θέμα αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον να επανεξετάσετε ή και να καταργήσετε ένα τέτοιο σύστημα. Και αυτό, ελπίζω να μην σας πειράζει, που το λέω, ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη δαπανούν τις κοινοτικέ πιστώσεις. Και οι 28 κυβερνήσεις ενδιαφέρονται να δαπανίσουν όλες τις πιστώσεις του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και δεν συζητιέται μετά ποια προστιθέμενη αξία ε, επιφέρει αυτή η ενωσιακή χρηματοδότηση για τους πολίτες. Αυτό ισχύει για την Ολλανδία. Να τα ξαναδούμε λοιπόν αυτά τα συστήματα για να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση των δημοσίων πόρων. Και ένα δεύτερο που νομίζω ότι έχετε βαρεθεί να με ακούτε να το λέω είναι καλύτερη ενημέρωση. Καλύτερη ενημέρωση για το πώς, για το πώς δαπανώνται οι δημόσιες δαπάνες. Τα τελευταία χρόνια που είμαι μέλος του ελεκτικού συνεδρίου στην Ολλανδία ορισμένες φορές εκπλήσωμαι από την έλλειψη Καλή ενημέρωση για το πώ δαπανήθηκαν δημόσιε δαπάνε. Εάν δεν έχουμε πληροφορίε για αυτά, για το τι επιπτώσει έχουν στην κοινωνία οι δαπάνε αυτέ. δεν μπορούμε να τα βελτιώσουμε μετά. Δεν έχουμε δηλαδή μια δυνατότητα να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Εάν δεν γίνονται σωστέ αποτιμήσει το πώ έχουν δαπανηθεί. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωση των δημοσίων δαπανών από αυτήν την πλευρά. Περισσότερη ενημέρωση. Και επίση να έχουμε και ε, ανοιχτή ανταλλαγή δεδομένων ούτως ώστε να εμπλακούν και οι επιχειρήσεις και το κοινό για να μάθουν πρώτα απ' όλα πώς δαπανώνται τα χρήματά τους. Νομίζω ότι έτσι θα αυξηθεί με δραματικό τρόπο η αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Βαλερή Ραμπού. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σταθώ στο διαστρωτικό έλλειμμα και πάλι, διότι υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις από αυτού. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θα μπορούσαμε να έχουμε σε μια ιστοσελίδα αναχώρα τους βασικούς δείκτες, δηλαδή στόχος για το διαρθρωτικό έλλειμμα και τις συνέπειες οποιασδήποτε μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος στην ανάπτυξη και ή τις επενδύσεις. Διότι νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται τι είναι η ανάπτυξη, όλοι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει συνέπειες στην ανάπτυξη έστω ότι μειώνουμε το διαρθρωτικό έλλειμμα κατά 0,1% ή 0,2%. Ποιες είναι οι συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη αναχώρα. Ποιες είναι οι συνέπειες για τις επενδύσεις αναχώρα. Έτσι ώστε ο καθής να μπορεί να καταλάβει ποιες είναι οι συνέπειες οποιασδήποτε μείωσης ε, στο διαρθρωτικό έλλειμμα θεωρώ ότι θα ήταν ουσιαστικό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι φέρπει ε, σε αυτή τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, κυρίως μέσω του διαρθρωτικού ελλείμματος. Μια δεύτερη πρόταση που θα ήθελα να κάνω είναι πώς, και εδώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας, όταν σχεδιάζεται μια δημόσια πολιτική, όταν γίνεται μια αξιολόγηση από αυτής της πολιτικής. Πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά με το θεματολόγιο 2020. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι γίνεται το τάδε στη Γαλλία, γίνεται το τάδε στην Ιταλία, το δίνα στις κάτω χώρες. Πώς σχετίζονται αυτά με το θεματολόγιο 2020 και ποια είναι η προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να επιφέρει όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι με αυτές τις δύο ιδέες, με αυτές τις δύο προτάσεις, τη μία για τον τρόπο ε, που διαχειριζόμαστε τη δημόσια οικονομικά και τα άλλα ως προς τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές στις χώρες μας που ε, καταρτίζονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το πώς σχετίζονται αυτά με το θεματολόγιο 2020, και κάθε φορά που κάνουμε κάτι ή προσαρμόζουμε το διαρθρωτικό έλλειμμα, τι συνέπειες έχει αυτό για την οικονομική ανάπτυξη, τι συνέπειες έχει αυτό για τις επενδύσεις, τι συνέπειες έχει αυτό για τις θέσεις εργασίας. Θεωρώ ότι θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για όλους και σίγουρα για τους πολίτες, εάν μπορέσουμε να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες σαφώς. Ευχαριστώ πολύ. απαντήσω κι εγώ σε μια γενική ερώτηση από το Βελγικό Κοινοβούλιο που ακούσαμε. Είναι κάτι γενικό, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Ντάσελβλουμ ότι πρέπει να έχουμε μια σταδιακή προσέγγιση. Συμφωνώ. Γιατί με άσπρο μαύρο δεν προχωράμε. Ιδεοδός, όπως είπα, ένας υπουργό οικονομικών της Ευρωζώνης θα είχε νόημα. Ένας υπουργό οικονομικών τι κάνει, ελέγχει τον εθνικό προπολογισμό. Σε ένα ε, στο ομοσπονδιακό κράτος υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια στα επιμέρους κρατήδια. Λοιπόν, δεν λέω όμως ότι αυτό θα γίνει σύντομα, αλλά σίγουρα πρέπει να βρούμε τρόπο να βελτιώσουμε το σύστημά μας. Και από αυτό που ακούσαμε, κατά τη γνώμη μου, από τη μια μεριά ο σημερινός μηχανισμός δεν είναι βέλτιστος, αλλά όχι αναποτελεσματικός, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει και των σχολείων και των νησιών που εκφράζονται. Υπάρχει λοιπόν αυτό το περιθώριο βελτίωσης και αυτό πρέπει να συνδυαστεί και είναι κεντρική σημασία πώς θα συνδυάσουμε το θέμα αυτό του ενστερισμού, πώς δηλαδή δεν θα υπάρξει αναρχία, αλλά οι χώρες θα υιοθετούν τα μέτρα, αλλά και θα τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά. Θα μπορούσαν οι κανόνες να εξελιχθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ έρχομαι στο θέμα της ευελιξίας. Θα μπορούσαμε κάλλιστα, αν θέλαμε, να λάβουμε υπόψη μας έκτακτες συνθήκες που δεν ελέγχονται από τις χώρες μέλη, όπως το προσφυγικό. Επιτρέπεται, δεν απαγορεύεται από τους κανόνες και να λάβουμε υπόψη μας μια διαστρωτική μεταρρύθμιση όσον αφορά τους μακροχρόνιους στόχους και να μην λάβουμε απόψη, υπόψη μας την συγχρηματοδότηση, κάποια στοιχεία του διαφορετικού ελλείμματο. Εντάξει, υπάρχουν περιθώρια, μπορεί να είναι στενά και με περιορισμού, αλλά συμφωνώ απόλυτα με το Συμβούλιο που είπε αυτό μπορεί να γίνει για ένα χρόνο, μόνο για ένα χρόνο. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο βελτίωση για την εφαρμογή τη ευελιξία, αλλά υπάρχει και περιθώριο για το πώ θα εφαρμόσουμε καλύτερα το σύμφωνο σταθερότητα. Και αυτά που είπατε για το διορθωτικό έλλειμμα είναι ζωτική σημασία. Πρέπει να αναλύσουμε όχι μόνο πώς διαμορφώνεται, αλλά και πώς υπολογίζεται. Μερικές φορές υπάρχουν αποτελέσματα σε αυτά που δεν είναι απόλυτα λογικά. Η χώρα που ξέρω εγώ καλύτερα, βάσει αυτού του μαθηματικού τύπου, δεν θα έπρεπε να αναπτυχθεί. Αν αναπτυχθεί λοιπόν 1%, ακόμα και αν δεν αυξηθεί σε ονομαστικές τιμές, φαίνεται σαν μείωση του διαφορετικού ελλείμματος. Γιατί, γιατί οι υπολογισμοί έλεγαν όχι, δεν θα αναπτυχθείτε. Αν αναπτυχθείτε παραβιάζετε τους κανόνες. Ε, προφανώς δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνουν κατανοητές οι ρυθμίσεις μας. Αυτά νομίζω συζητούν και στο Εθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε ο ονομαστικός χαρακτήρας να λυθεί περισσότερο υπόψη χωρίς να λέμε ότι πρέπει να απαλλαγούμε πλήρως από την διαρθρωτική προσέγγιση. Συνεπώς, υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις και ο συνδυασμός εθνικής και ευρωπαϊκής αποδοχής και λογοδοσίας αποτελεί στοιχείο κλειδί. Συνεπώς η σημερινή συζήτηση ήταν πολύ συγκεκριμένη και αποτελεσματική. Είναι καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τέλος ο συμπρόεδρος. Ωραία, ας μην συνεχίσουμε τα συγχαρητήρια των προς τον άλλον. Εγώ συγχαρητήρια σε εσά θέλω να δώσω για τον τρόπο που ηγηθήκατε τη συζήτηση αυτής. Έχουμε διάλειμμα για καφέ. Ένα τέταρτο. Έχουμε αργήσει ήδη. Τα κύρια ζητήματα έχουν τεθεί πάντως. Ευχαριστώ πολύ και θα ξαναβρεθούμε εδώ στις 11.30. Και θα πάμε στον πρώτο όροφο στην αίθουσα Γεγουντή Μενουίν. Ευχαριστώ πολύ.